I think we can start a little bit later. Ας αρχίσουμε, νομίζω ότι έχει κάπως βέβαια ε, προχωρήσει η ώρα. Σας καλωσορίζω στο, στη συνεδρίασή μας. Ε, ε πως έχετε ενστάσεις για την ημερησία διάταξη. Αν όχι, τότε να εγκρίνουμε το πρακτικό της 28ης Πέμπτου δεν υπάρχουν παρατηρήσεις. Ανακοινώσεις του Πρόεδρου ακόμη δεν έχουμε. Προχωράμε στο υπαριθμό 4. Καλώς ήρθατε κύριε Ζωζέ Μανουέλ Φερνάντες που είστε εισηγητής για τον προπολογισμό 2016, της Επιτροπής Προπολογισμών δηλαδή. Καλώς ήρθατε εδώ στην Επιτροπή Μεταφορών. Ευτυχώς που το αεροπλάνο σας δεν άργησε γιατί αλλιώς θα αισθανόμασταν κάποια ε, ιδιαίτερη στενοχώρια. Έχουμε μια καλή συνεργασία παραδοσιακά ανάμεσα στις δύο επιτροπές, δηλαδή Προπολογισμών και Μεταφορών, είναι σημαντικό οι προτεραιότητε του Κοινοβουλίου να ληφθούν σοβαρά υπόψη από το Συμβούλιο σε ό,τι αφορά τον προπολογισμό και στον τομέα των μεταφορών, όχι βέβαια μόνο. Και αυτό χρειάζεται να έχουμε μια κοινή γραμμή. Σα υπενθυμίζω ότι έχουμε και τι ε, διαπραγματεύσει που πρέπει να εφαρμόσουμε για τον ΕΦΣΥ. Σα παρακαλώ κύριε Φερνάντε, πέστε λίγα λόγια τώρα για την διαδικασία του προπολογισμού. Έχετε το λόγο, αγαπητοί Ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση. Λόγω <clears throat> των μεταφορών, όχι των δικών σας βέβαια. Καθυστέρηση πτήση μου. Ήδη έχουμε υιοθετήσει τις προτεραιότητες μας, για τις κατευθυντήριες γραμμές μιλάω, τα τρία ε που λέμε στα γαλλικά, επιχειρήσεις απασχόληση, επιχειρηματικότητα και εσωτερική αλληλεγγύη και εξωτερική αλληλεγγύη. Δεν μπορούμε εμείς να αγνοήσουμε το τι συμβαίνει εκτός Ένωσης και φυσικά ασφάλεια. Αυτές οι προτεραιότητες έχουν συνέπειες και θα μπορούσαν εν μέρη να βοηθήσουν την απασχόληση και σε σχέση με την απασχόληση φυσικά έχουμε πολλά σχέδια. Βασιζόμαστε στην ιδέα ότι οι υποχρεώσεις θα γίνουν σεβαστές. Και αυτό ισχύει για όλα τα όργανα. Αλλά είναι και μια παρατήρηση προς το Συμβούλιο άμεσα την κάνουμε. Όταν λέμε ότι πρέπει να γίνουν σεβαστές οι υποχρεώσεις, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να γίνουν ε, σεβαστές οι πληρωμές. Οι πληρωμές είναι η λογική συνέπεια των πιστώσεων υποχρεώσεων. Όταν μιλάμε για προβλήματα πληρωμών, μιλάμε για προβλήματα με τα προαποφασισμένα, με τους ε, λογαριασμούς τους οποίους είμαστε υποχρεωμένοι να πληρώσουμε. Και μιλάμε επίσης για θέματα αξιοπιστίας. Είναι ντροπή είναι απαράδεκτο το Συμβούλιο να μην ε, διαθέτει τα χρήματα της πιστώσης που απαιτούνται ε, και είναι συνέπεια των δηλώσεών του και συνέπεια των πιστώσεων υποχρεώσεων που έχουν ήδη γίνει δεκτές. Μιλάμε για το νέο δημοσιονομικό πολιετές. Μέσα σε αυτό υπάρχει μια κάποια ευελιξία. Υπάρχουν τα λεγόμενα μέσα ευελιξίας και υπάρχει και το σφαιρικό λεγόμενο περιθώριο, το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε από το 2016. Και οι υποχρεώσεις από τα προηγούμενα χρόνια μπορούν να καλυφθούν από συγκεκριμένες πολιτικές προτεραιότητες με στόχο την ανάπτυξη και την απασχόληση. Εμείς θέλουμε λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε αυτή την ευελιξία και γι' αυτό αποδεχθήκαμε έναν προϋπολογισμό χαμηλότερο, ένα πολυετές πλαίσιο χαμηλότερο σε σχέση με το προηγούμενο 7-13 και είναι φυσικό ότι στα πλαίσια της συζήτησης για το προϋπολογισμό πλέον σήμερα τίθεται το θέμα των υποχρεώσεων στις οποίες έχουμε καταλήξει για το ΕΦΣΥ και για το Horizon 2020 και για το Connecting Europe. Επ' αυτών έχουμε τους ίδιους στόχους που είχαμε και κατά τη διάρκεια των πρώτων διαπραγματεύσεων και ευχαριστώ τους δύο εισηγητές σας που με είχαν βοηθήσει να καταλήξουμε σε ένα αποτέλεσμα που είναι καλό αλλά δεν τέλειωσε η δουλειά μας εδώ. Ο στόχος παραμένει, όπως έχω επανειλημμένα πει, στόχος ελαχιστοποίησης όσο περισσότερο γίνεται των επιπτώσεων των προτάσεων αυτών για το Horizon 2020. Είναι ξεκάθαρο και σε επίπεδο κανονισμού και πολιτικά ότι σε κάθε δημοσιονομική διαδικασία θα έχουμε ανάγκη και από εσά φυσικά, από τη δική σας επιτροπή, ε, να επιδιώξουμε τον στόχο, επαναλαμβάνω, της μείωσης της, ε, των αρνητικών συνεπειών επί του Connecting Europe και του Horizon 2020. Για το χρονοδιάγραμμα τώρα, να θυμίσω ότι στις 27 Μαΐου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε την τελική πρόταση για το σχέδιο προϋπολογισμού. Θυμίζω ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία βέβαια, το Συμβούλιο θα αναγνώσει σε εισαγωγικά την πρόταση, το ίδιο θα κάνουμε και εμείς, θα εξετάσουμε την πρόταση και θα προσπαθήσουμε να δούμε αν είναι συμβατή η πρόταση της Επιτροπής και με τις δικές μας προτεραιότητες. Επί το περιθωρίου έχουμε ένα περιορισμένο περιθώριο, ιδιαίτερα στο 1, μόνο 200 εκατομμύρια. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα σε πιλωτικά προγράμματα, αλλά Μέχρι την 3η Σεπτεμβρίου προθεσμία κατάθεσης των τροπολογιών που θα εξεταχθούν στο Στρασβούργο στις 23 Σεπτεμβρίου και θα εξεταστεί αυτά στην Αρμόδια Επιτροπή και τον Οκτώβριο θα ψηφίσουμε στον προϋπολογισμό στην Ολομέλεια. Έχουμε μετά από τις 28 Οκτωβρίου μέχρι τις 19 Νοεμβρίου τη διαδικασία συνδιαλλαγής. Όπως είπα, στο σχέδιο προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν έχουμε καταλήξει για το ΕΦΣΥ. Θα απαιτηθεί μια διορθωτική δημοσιονομική επιστολή. είχε προβλεφθεί εδώ μία αύξηση 43% στις υποχρεώσεις, αλλά δεν είχαμε ακόμα τότε τις επιπτώσεις, τις μειώσεις που θα προκαλούσε στο ΕΦΣΥ. Συνολικά για τον προϋπολογισμό 37,9 στις υποχρεώσεις σε σχέση με το 15 Μιλάω πάντα για το σχέδιο της Επιτροπής και 18,9 στις πληρωμές για τις εξωτερικές υπηρεσίε. Συνολικά. Σφαιρικά. Δεν μπορεί να υπάρξει μία μείωση 5% όπως έχει προταθεί. Εξίσου για όλες τις εξωτερικές υπηρεσίες όλες. Για την ΕΑΣΑ, την ασφάλεια την αεροπορική, υπάρχει μια πολύ μικρή μείωση κατά 0,8%. Μια μικρή αύξηση 0,2% για τα φάρμακα για τους σιδηροδρόμους έχουμε μια ελάχιστη αύξηση 0,35. Ε, λοιπόν, το περιθώριο στον τίτλο 1α είναι μικρό. 100 εκατομμύρια λέει το ο Μετά από την ανάγνωση του Συμβουλίου και μετά τις προτάσεις του Συμβουλίου τότε θα έλθει η σειρά των τροπολογιών μας. Εγώ ήρθα εδώ σήμερα για να σας ακούσω κυρίως. Ήρθα εδώ σήμερα για να συλλέξω τις δικές σας προτεραιότητες που είναι σημαντικές και για τις κατευθυντήριες γραμμές τις οποίες αναφέρθηκα και για να προσπαθήσουμε μαζί να φτιάξουμε τον καλύτερο δυνατό προϋπολογισμό. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσετε. Ευχαριστώ πολύ αγαπητέ ε, Φερνάντες. αναμένεται όλη την συζήτηση. Πριν δώσω τώρα τον λόγο στον κύριο Σαλίνη, εισηγητή προϋπολογισμού της ομάδας μεταφορών. Καλωσορίζω ομάδα 15 φοιτητών από την Σορβόνη ε, που σπουδάζουν αντικείμενο σχετικό με τι μεταφορές. Καλώς ήρθατε στην Επιτροπή μας. Τώρα θα δώσω το λόγο στον Μάσιμο Μασιμιλιάνο, με συγχωρείτε Σαντίνη. Και μας. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Φερνάντες για την συνοπτική παρουσίαση της μεθόδου εργασίας την οποία υιοθέτησε και υπενθύμησε τις προτεραιότητες επί, των οποίων εξελίσσεται θα έλεγα η διαδικασία για την οικοδόμηση του προϋπολογισμού του 16 στα θέματα που μας ενδιαφέρει. Εμείς έχουμε μια μεγάλη ανησυχία όπως είναι γνωστό και το απέδειξαν οι διαπραγματεύσεις μια ανησυχία για την σχέση ε, με, ανάμεσα στο Connecting Europe, στο ΕΦΣΥ, και στο νέο πρόγραμμα του Juncker. Είναι μια καινοτομία και δεν θα πρέπει να φυγεί η ανεξαρτησία του Connecting Europe το οποίο στηρίζει επενδυτικές διδανότητες ε, πολύ σημαντικές. Ένα κλασικό παράδειγμα. Οι λιγότερο ενδιαφέρουσες για τους ιδιώτες επενδυτές μορφές επενδύσεων οι οποίες θα φυγούν εν πολλής από τη νέα μορφή που προβλέπεται στο εσωτερικό του ΕΣΥ για την χρηματοδότηση. Δηλαδή οι κανόνες στην ουσία οδηγούν σε σενάρια τα οποία επενδύσεις στον τομέα των σιδηροδρόμων ή των παραποτάμιων συγκοινωνιών κτλ. γίνονται πολύ περίπλοκες και λιγότερο ενδιαφέρουσες και συμφέρουσες. Το πρώτο μεγάλο λοιπόν ερώτημα το οποίο τίθεται είναι μετά από αυτά που είπατε <clears throat> για το περιθώριο είναι να υπάρξει μια κάποια διαφάνεια για το πόσο από το περιθώριο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε έτσι ώστε η μείωση του ΣΕΦ να μην οδηγήσει σε αρνητικές επιπτώσεις. Τι περιθώριο δηλαδή είναι αυτό το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για αντιστάθμιση των μειώσεων. Δεν στέκομαι τώρα σε όλα τα υπόλοιπα θέματα τα οποία φύγουν τις ανησυχίες μας για τον προϋπολογισμό. Θα σας τα θυμίσω λίγο συνοπτικά. Είπατε και εσείς την ανάγκη που υπάρχει για μια χρήσιμη παρέμβαση στις εξωτερικές υπηρεσίες και για το τέταρτο σιδηροδρομικό πακέτο. Ελπίζουμε ότι οι εθνικές υπηρεσίες να συνδυάζονται με την ευρωπαϊκή έτσι ώστε να έχουν τα πλαίσια λειτουργίας του στην εμβέλεια που απαιτείται. Ο ΕΝΙΕ, e η Ευρωπαϊκή Ουρανή, απαραίτητες επενδύσεις για την ασφάλεια των επιβατών, φυσικά των αερομεταφορών, τα συμφέροντα των ταξιδιωτών, να μην θεωρούνται οι αερομεταφορές σαν απλό μέσο διασύνδεσης των υποδομών στην Ευρώπη, αλλά σαν κίνητρο και για την ανάκαμψη των εσωτερικών αγορών. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια σύνδεση ανάμεσα στην ανάπτυξη και τις, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις στις αερομεταφορές. Αυτό όμως αφορά την επόμενη φάση των εργασιών. Ξέρετε ότι σήμερα η μισή από τους κατοίκους του κόσμου ζουν σε αστικές περιοχές και τίθεται και θέμα φυσικά η φορεία των μεταφορών, δεν το αγνοούμε αυτό. Υπάρχουν πολλά θέματα όπως είπατε που πρέπει να μας απασχολήσουν. Αλλά το βασικό είναι η σχέση ανάμεσα στο τσεφ και το ΕΦΣΙ και το τσεφ συγγνώμη και η σχέση ανάμεσα στο ΕΦΣΙ και το Horizon 2020. Ευχαριστώ. Πυρίνσκι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμη κύριε Ισηγητά και εσείς κυρίες και κύριοι, συμφωνώ με την τελευταία σας δήλωση σε ό,τι αφορά τον προϋπολογισμό για τις μεταφορές όπου η κινητικότητα είναι από τους πιο σημαντικούς παράγοντες ήδη για τον προϋπολογισμό του 2016 και είναι πολύ ευχάριστο που έχουμε την δυνατότητα να ανταλλάξουμε απόψεις και να εξετάσουμε τις προτεραιότητες. Ο τίτλος Mobility and Transport βλέπει μια αύξηση και στις πιστώσεις υποχρώσεων και στις πιστώσεις πληρωμών σε σχέση με το 2015. Είμαι βέβαιος ωστόσο ότι θα έχετε προσέξει κι εσείς ότι στα διάφορα μεμονωμένα άρθρα αναφύονται και μειώσεις, περικοπές είτε των υποχρώσεων είτε των πληρωμών. Και λιγότερες πιστώσεις πληρωμών σε σχέση με τις πιστώσεις υποχρεώσεων του 2015. Και εννοώ βέβαια για τη διευκόλυνση συνδέοντας την Ευρώπη και για την ασφάλεια των μεταφορών. Μπορεί αυτή η δυσκολία να προέρχεται από πολιετή προγράμματα και την κατανομή των κονδυλίων ανάμεσα σε παραπάνω από ένα χρόνο. Όμως πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην υποτιμήσουμε το ενδεχόμενο στο μέλλον να επανέλθει, να ξαναδούμε δηλαδή μια ανεπάρκεια κονδυλίων όπου συγκεντρώνονται πλήρω οι λογαριασμοί προ τα τέλη τη περίοδου. Τώρα, για την διευκόνηση συνδέοντα την Ευρώπη υπάρχει στις υποχρώσεις σημαντική αύξηση και κάποια μείωση στις πληρωμές. Μετά την έγκριση του κανονισμού ΕΦΣΥ θα προτείνει τροποποίηση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. στη έφευση. Ο ΕΦΣΥ περιλαμβάνει δήλωση ότι όλες, όλα τα κονδύλια για τα ταμεία εγγύσεων θα εγκρίνονται και από το Κοινοβούλιο και από το Συμβούλιο μέσα στα πλαίσια της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού και σε πλήρη συμμόρφωση με τις σχετικές διατάξεις του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020. Εν προκειμένου, θα ήθελα να κάνω την εξής ερώτηση. Μπορείτε εσείς κύριε Γκοντζάλες ή Φερνάντες, συγγνώμη, να Χρησιμοποιήστε την ευκαιρία που δίνουν οι αιτήσεις διαδικασίες προπολογισμών να αποκαταστήσετε τις πιστώσεις του ΣΥΕΦ στο μέγιστο δυνατό βαθμό και βλέπετε να υπάρχει δυνατότητα. Τώρα, για τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων, Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων, σας επισημαίνω ότι τα ποσά που προτείνεται να δοθούν στον οργανισμό αυτό και για το δημοσιονομικό αποθεματικό για το ERA. Το Κοινοβούλιο προέβησε καταρχήν συμφωνία όπου δίνει νέες αρμοδιότητες στον οργανισμό σιδηροδρόμων και το ερώτημα είναι αν θα υπάρχει επαρκής χρηματοδότηση του οργανισμού σιδηροδρόμων για την αντιμετώπιση των νέων καθηκόντων του και στην αρχική φάση όπου δεν θα εισπράττονται ακόμα τέλη και εισφορές και πώς μπορεί να διασφαλιστεί αυτό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και εν προκειμένου μου επισημάνθηκε μια δήλωση από τις υπηρεσίες της Κομισιόν για τους πόρους του οργανισμού που έχει ως εξής. Το πρώτο πακέτο σιδηροδρόμων δίνει στον οργανισμό νέες αρμοδιότητες. Για παράδειγμα, πιστοποιητικά και άδειες κυκλοφορίας για νέα οχήματα. Δεν αποκλείεται στην αρχική μεταβατική περίοδο να μην διατίθεται ακόμα, να μην λαμβάνονται, να μην εισπράττονται ακόμα τέλη και εισφορές, ενώ θα πρέπει να προσληφθεί κόσμος και να εκπαιδευτεί για να αποφευθεί οποιαδήποτε διακοπή λειτουργία της αγοράς των σιδηροδρόμων θα πράξουν πάνω δυνατόν η υπηρεσία της Κομισιόν για να ε, βάλουν σε αποθεματικό όσο το δυνατόν περισσότερα κονδύλια για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις καταστάσεις αυτές. Τώρα για τον τουρισμό. Δεν υπάρχει ειδικό κονδύλιο για τον τουρισμό. Τα σχετικά έργα μπορούν να ε, χρηματοδοτηθούν και από το πρόγραμμα COSME για τις μικρές και μεσές επιχειρήσεις γίνεται μείωση και υποχρώσεων και πληρωμών σε σχέση με το 2015 όπως γνωρίζουμε και εδώ θέλω να σας επισημάνω ιδίω. ότι υπάρχει μια προσδοκία σημαντική αγαπητέ Φερνάντες ότι θα δοθεί υποστήριξη σε προτινόμενα πιλωτικά προγράμματα και προπαρασκευαστικές δράσεις για τον τουρισμό που έχουν υποβληθεί ως προτάσεις δικές μας και θα ήθελα να σας προτρέψω και στο όνομα των συναδέλφων μου που ενδιαφέρονται πολύ για τα θέματα του τουρισμού να μας υποστηρίξετε. Ευχαριστώ. Τελίτσκα. Πάβελ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εκ μέρους του Ντομινίκ Ρικέ μιλάω, εκείνος χρειάστηκε να φύγει και λυπάται που δεν μπορεί να είναι παρόν στη συζήτηση αυτή. Ευχαρίστω όμως θα σας μεταφέρω τις παρατηρήσεις του. Να σας πω επίσης ότι συμφωνώ με περίπου όλα όσα λέξα, αλλά αλλιώς δεν θα μιλούσα εκ μέρους του. Κύριε Φερνάντες, αναφερθήκατε στο ότι θα μας ακούτε. Μπορώ να πω ότι πολλές από τις παρατηρήσεις είναι θετικές. Πρέπει να πούμε ότι στο δύσκολο πλαίσιο με το χρονοδιάγραμμα που έχουμε στη διάθεσή μας και ο Ντομινίκ και εγώ αλλά και η υπόλοιπη ομάδα νομίζω μπορεί να πει ότι έχετε κάνει πολύ καλή δουλειά και αξίζεται πραγματικά ιδιαίτερες ευχαριστίες. Επίσης εκτιμούμε όλους ιδιαίτερος το γεγονός ότι έχετε εξετάσει τα συμφέροντα της Επιτροπής αυτής και προσπαθείτε με τις προσπάθειές σας να βοηθήσετε στο βαθμό του εφικτού βέβαια στις συζητήσεις να ελαχιστοποιήσετε τις επιπτώσεις πάνω στο συνδέοντα στην Ευρώπη και στο Horizon 2020. Θα φτάσουμε βέβαια αργότερα τη χρονιά αυτή και το 2000, με τον προπολισμό το 2016 θα κληθούμε να δώσουμε νέα μάχη. Το σχέδιό σας Πάντως πιστεύουμε ότι είναι μια πολύ καλή βάση πράγματι. Κατά τη γνώμη μας αντικατοπτρίζει πλήρως τις ανησυχίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πιο συγκεκριμένα της δικιάς μας Επιτροπής. Τώρα, αναφερθήκατε στο Συμβούλιο. Είπατε ότι πρέπει κανείς να πληρώνει τους λογαριασμούς του και να σέβεται τις υποχρώσεις που αναλαμβάνει. Προσυπογράφω απόλυτα. Και νομίζω ότι θα έπρεπε εξ να δούμε τι έχει γίνει μέχρι τώρα και βάσει της εμπειρίας μας να προχωρήσουμε και να δώσουμε αργότερα μέσα στη χρονιά αυτή τη μάχη που θα κληθούμε να δώσουμε ανάλογα. Κατά τα άλλα, πρέπει να προσπαθήσουμε να μεγιστοποιήσουμε όσο γίνεται περισσότερο το περιθώριο που έχουμε από τον προπολογισμό. Αυτό είναι πολύ βασικό για να ενισχύσουμε τη στήριξή μας σε προγράμματα τα οποία αποτελούν ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, έργα υποδομών βασικά. Θα δούμε τελικά ποιες θα είναι οι προτάσεις οι οποίες θα γίνουν και στο συνδέοντας την Ευρώπη. Και όταν θα έχουμε κάτι πιο συγκεκριμένο, θα ξέρουμε τι ποσό θα πάει εκεί και τι μένει στο περιθώριο. Πάντως φοβάμαι ότι τα ποσά είναι επιβεβαίωση των προσδοκιών μας. τριπλασιάζοντας τον προπολογισμό μπορούμε να δαπανίσουμε. Τώρα έρχομαι στους διάφορους οργανισμούς. Ο Ντομινίκ θέλει να υπογραμμίσει ότι συμφωνεί με το ότι κάθε οργανισμό πρέπει να τον εξετάζουμε διαφορετικά. Το είπε αυτό και ο προλαλή αλλά και ο εισηγητής. Και ο και ο Έχουμε και κάποια καινούργια κατάσταση. Εδώ θα ήθελα να αναφερθώ στον Οργανισμό για την Ασφάλεια Αεροπορίας, για παράδειγμα, και στον Οργανισμό Σιδηροδρόμων, που ασχολείται με την αδειοδότηση και κυρίως το RTMS, που πάνω σε αυτό πρέπει να επικεντρωθούμε. Τώρα, εκ μέρους του Ντομινίκ, θέλω να επιστήσω στην προσοχή σας και κάτι πιο συγκεκριμένο. Πρωτοβουλίες τεχνολογικής φύσης που είναι αναγκαίες για την ανταγωνιστικότητα των μεταφορών στην Ευρώπη. Μετά τις διαπραγματεύσεις για το ΕΦΣΥ, το Ευρωπαϊκό Αυτό Ταμείο, μιλάμε για 5 δισεκατομμύρια. Το ΣΥΖΑΣ δύο φορές υπολογίζεται φέτος. Μέσω του συνδέοντας την Ευρώπη πρώτον και δεύτερον μέσω του Horizon 2020 όταν η ενιαία εθέρεση ήταν, είναι περισσότερο αναγκαία από ποτέ. Κάτι πολύ ανησυχητικό αν μη τι άλλο. Τέλος, shift to rail, η μεταφορά δηλαδή στις δρομικές μεταφορές θα επηρεστεί από την μείωση του Horizon 2020. Γι' αυτό θέλω να σας εκφράσω εδώ τις ανησυχίες του Ντομινίκ επ' αυτού ότι παρόλο που η κοινοπραξία εγκρίθηκε πέρυσι, έχουν υπάρξει καθυστερήσεις όσον αφορά την έγκριση των υποχρεώσεων. Το σχέδιο έκθεσης πάντως εντοπίζει με σαφήνεια το τι θα αντιμετωπίσουμε. Για άλλη μια φορά, είναι μια καλή προσπάθεια. Αν θέλετε τη στήριξη της Επιτροπής μας, δεν μπορώ βέβαια να μιλήσω εκ μέρους όλης της Επιτροπής, αλλά εκ μέρους του Άλντε, να ξέρετε ότι θα έχετε τη στήριξή μας, προκειμένου να πετύχετε όσο γίνεται περισσότερα θετικά αποτελέσματα και να μειώσετε όσο γίνεται περισσότερα εκείνα τα οποία θα είναι αρνητικά στο Συμβούλιο. Πάντως πρέπει να το αναγνωρίσουμε στην Επιτροπή μας ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιούργησε ένα καλό δίδυμο με το Συμβούλιο. Πρέπει να το δεχτούμε αυτό. Θα έχετε τη στήριξή μας. Ευχαριστώ. Ο πρόεδρος, ο πρόεδρος Κράμερ, η κυρία Καρυμάντελη. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Σιγητά, θα είμαι πολύ συγκεκριμένη. Πρέπει να κάνουμε διάκριση στα πειραματικά προγράμματα και τις προπαρασκευαστικές δράσεις. Εμείς έχουμε κάνει συγκεκριμένες προτάσεις για προπαρασκευαστικές δράσεις όσον αφορά τα νυχτερινά τρένα. 980.000 ευρώ έχουμε δώσει μόνο. Πού βρισκόμαστε σήμερα από αυτού. Δεύτερον, οι αποφάσεις, τα διάφορα συμπεράσματα από την Επιτροπή Τραν υπογραμμίζουν ότι υπάρχουν κατά προτεραιότητα γραμμές. Και θέλω να ξέρω ποια είναι η ημερομηνία που προβλέπετε για την επιλογή. 31η Αυγούστου. Πού ακριβώς βρισκόμαστε σήμερα. Επίσης, κύριε Σιγητά, θέλω να σας πω και κάτι ακόμα. Δεν κατάλαβα καλά ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα και δεν κατάλαβα καλά ποιο είναι το πλαίσιο αρχής που θα εφαρμόσετε σε αυτήν τη δημοσιονομική διαδικασία. Γνωρίζουμε ότι σήμερα ο μηχανισμός της διασύνδεσης, ένα μέρος πάει στο σχέδιο Juncker, αλλά συγκεκριμένα μπορείτε εσείς να μας πείτε ποιες θα είναι οι συνέπειες για τα προγράμματα εκείνα τα οποία δεν θα προχωρήσουν μας μιλάτε για έναν τομέα ε, για τον οποίο αναφερόμαστε όλο και πιο στην Επιτροπή μας, που είναι ο βιώσιμος τουρισμός. Ποιο πλαίσιο εσείς θα θεσπίσετε όταν μιλάμε για προγράμματα κόσμου. Έχουμε απαντήσεις συγκεκριμένες και μπορούμε να έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα έτσι ώστε μακροπρόθεσμα να ξέρουμε πότε θα γίνει τι. Ευχαριστώ. έχω σημειώσει και το δικό όνομα στον κατάλογο των αγορητών. Πρώτα ο Κόξ είπε ότι οι σιδηρόδρομοι στην Ευρώπη είναι σαν password και τα κενά εντοπίζονται εκεί όπου είναι τα σύνορα. Παρόλο που έχουμε τα τελευταία 20 χρόνια δαπανίσει δισεκατομμύρια, δεν τα καταφέραμε να ολοκληρωθούν τα δίκτυα. Έχετε κάποια ιδέα πώς μπορείτε να δώσετε προτεραιότητα σε ορισμένα έργα από την πλευρά, από την, την της Επιτροπής έτσι ώστε οι χώρες μέλη να μην παίρνουν χρήματα από τον προϋπολογισμό μονάχα για υλοποίηση δικών τους έργων εθνικών, αλλά και για υλοποίηση έργων κοινοτικού ενδιαφέροντος. Σε όλες τις παρατηρήσεις, τις παρατηρήσεις για τον FC υπάρχει μονάχα ένα έργο τέτοιο. Έτσι μου είπαν. Τώρα, Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εμείς εκπλαγήκαμε λίγο, ή πάντως δεν διασκεδάσαμε διόλου, για την κατάσταση Τη επιτροπή Προπολογισμών πέρσι. Διότι εμείς στην Επιτροπή μας είχαμε αποφασίσει ότι θα αφήσουμε, θα διατηρήσουμε τις ε, δημοσιονομικές, του δημοσιονομικούς όρους. Επειδή έχουμε τώρα λίγους ποδηλατοδρόμους, είχαμε πει 0,5% του προϋπολογισμού να πάνε στις, ε, στο πρόγραμμα Ευρωβελό και τα απέρριψε αυτά η Επιτροπή Προπολογισμών. Κοιτάξτε, καταλαβαίνω βέβαια ότι αυτό που σας ενδιαφέρει είναι να είναι θεσπισμένο το πλαίσιο. Εμείς όμως το πλαίσιο δεν το αλλάξαμε. Βάλαμε ορισμένε προτεραιότητε, ορισμένα κέντρα βάρου. Και εκεί η Επιτροπή Προπολογισμών έρχεται και λέει ότι αυτά τα κέντρα βάρου τη Επιτροπή Μεταφορών δεν μα ενδιαφέρουν, δεν τα αποδεχόμαστε. Αυτό κάπω μα φάνηκε παράδοξο. Αν ήσασταν μέλο και εσεί σε μια εξειδικευμένη κοινοβουλευτική επιτροπή, με τον ίδιο τρόπο θα αντιδρούσατε. Πώς είναι λοιπόν αυτό, έχετε κάποια ιδέα και στο μέλλον θα μπορέσετε να ταχθείτε υπέρ του σεβασμού και της στήρησης των ε, παρατηρήσεων των άλλων κοινοβουλευτικών επιτροπών. Τώρα, θα δώσω το λόγο κατεξαίρεση στον κύριο Κάμπ, ο οποίος τον ζήτησε εκτός ε, καταλόγου. Πρόεδρε, Θέλω να σας ευχαριστήσω γονατιστός που μου δίνετε το λόγο. Ναι, εντάξει. Ναι, πραγματικά σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Χαίρομαι πολύ που ο εισηγητής για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αγγίσεων, ο κ. Φερνάντες με τον κ. Μπούλμαν, ο κ. Φερνάντες είναι και εισηγητής για τον προπολογισμό 2016. Είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία για να ελέγξουμε κατά πόσο οι συμφωνίες που έχουμε πετύχει για το συνδέοντα στην Ευρώπη και το Ταμείο Αυτοεγγύσεων τελικά θα λειτουργήσουν καλά. Τα είπανε και ο Σαλίνη και οι των ε, Σοσιαλιστών ότι το βασικό είναι η απόδειξη. Περιμένουμε δηλαδή να δούμε συγκεκριμένα τα στοιχεία. Δεν ξέρουμε αν είναι καλό το γλυκό παρά μόνο όταν το φάμε. Θέλω λοιπόν να δω πόσο θα συνεισφέρει το ΣΕΦ και πόσα θα μπορέσουμε να πάρουμε πίσω από το περιθώριο το 2016. Τότε μόνο θα είναι σαφές για μας το πράγμα. Όσον αφορά τώρα τις ε, τεχνικές συμφωνίες για το πακέτο σιδηροδρόμων και ο κύριος Σαλίνη και άλλοι είπαν ότι πρέπει να χρηματοδοτεί κατάλληλα ο οργανισμός σιδηροδρόμων. Εγώ τώρα θα ήθελα περισσότερα χρήματα στην έρευνα, στον Horizon δηλαδή, για τις μεταφορές. Η έρευνα για την υγεία είναι πολύ σημαντική βέβαια, αλλά και η έρευνα για τις μεταφορές είναι πάρα μα πάρα πολύ σημαντική. Πρέπει να κάνουμε λοιπόν μια έκκληση για τα χρήματα αυτά στο Horizon 2020. Αυτό ήθελα να πω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Φερνάντες τώρα. Παρακαλώ κύριε Φερνάντες. Je vous remercie. Je remercie tous euh, les commentaires. Ευχαριστώ πολύ για τα σχόλια. Θα προσπαθήσω να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Μερικές ήταν παρόμοιες μεταξύ τους. Και θέλω να υπενθυμίσω ότι ο προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ένας μικρός προπολογισμό 1% του, του ΕΠ, του εχώριου. ...145 δισεκατομμύρια σε υποχρεώσεις. Αν θέλουμε να το συγκρίνουμε με τις Ηνωμένε Πολιτείες, εκεί είναι 20% του ΕΠ ο Ομοσπονδιακό προπολογισμό στι Ηνωμένε Πολιτείε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η αξία του είναι μεγάλη. Και πρέπει να το επαναλάβουμε ότι ο προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση 94% πάει στι επενδύσει. Μόνο 6% του προπολογισμού πηγαίνει στι διοικητικέ δαπάνε και στι λειτουργικέ δαπάνε. Τα στοιχεία αυτά λοιπόν δείχνουν πολύ καθαρά την προστεθέμενη αξία του προπολογισμού που σε πολλές χώρες είναι πάνω από το 50% σε επενδύσεις. Πρέπει επίσης να υπενθυμίσουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ένας βραχίωνας του προπολογισμού. Είμαστε νομοθετική εξουσία την εκτέλεση όμως του προπολογισμού την αναλαμβάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Φυσικά πρέπει να τηρούμε τους κανόνες και θα κάνω τα πάντα για την Επιτροπή Μεταφορών. Πρέπει να ξέρετε ότι αγωνίστηκα πάρα πολύ, σαν να ήμουν ένας από εσά. Έκανα ό,τι μπορούσα ως εισηγητής και υπάρχει ένα σημαντικό προηγούμενο και αυτό είναι η χρήση των μη χρησιμοποιημένων ήδη περιθωρίων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είχε καν μιλήσει γι' αυτό. Το κάναμε όμως. Και δείξαμε ότι σε κάθε δημοσιονομική διαδικασία, διαδικασία του προπολογισμού, θα έχουμε το Ταμείο Εγγύσεων. Πάντως υπάρχουν κανόνες που πρέπει να τηρούνται και ένας από τους κανόνες αυτούς, και εδώ απαντάω στον πρόεδρο, είναι η αρχή της οικουμενικότητας. Δηλαδή ότι δεν μπορούμε να βάζουμε ποσοστώσεις, δεν μπορούμε να κάνουμε earmarking, δεν επιτρέπεται αυτό, δεν είναι νόμιμο. Δεν μπορούμε να πούμε 5% για αυτό το πρόγραμμα κτλ. Και νομίζω ότι ακριβώς για αυτό το λόγο μια σημαντική σας ανησυχία δεν καθησυχάστηκε τελικά γιατί δεν το δέχτηκε αυτό η Επιτροπή Προπολογισμών που ζητούσατε. Τώρα, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο επενδύσεων. Το έφυση. Πρέπει να δούμε τι έργα θα προκριθούν τελικά. Πρόκειται για μια πρόκληση. Για μια ευκαιρία αλλά και μια πρόκληση. Τι λέει το, λέει είμαι εδώ για να χρηματοδοτήσω προγράμματα τα οποία δεν χρηματοδοτούνται από άλλα προγράμματα, ούτε από τα ταμεία, ούτε από τις οικονομικές αγορές. Ε, εγώ είμαι εδώ, αυτό το ταμείο, για να χρηματοδοτήσω βιώσιμα προγράμματα, τα οποία σέβονται τη στρατηγική 2020. Αλλά δεν είναι θεματικά ούτε γεωγραφικά. Είναι λοιπόν μια πρόκληση για τους δικαιούχους. Είναι μια πρόκληση για την έρευνα. Είναι μια πρόκληση για τις μεταφορές. Είναι μια πρόκληση για τον τουρισμό. Και ο τουρισμός είναι μία δυνατότητα χρηματοδότησης. Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής, η προτεραιότητα των μεταφορών υπάρχει στην έκθεση. Δεν μπορεί βέβαια κανείς να πει από τώρα ποια θα είναι τα προγράμματα που θα χρηματοδοτηθούν, γιατί αυτό θα εξαρτηθεί από τον ενδιαφέρον που θα δείξουν οι ενδιαφερόμενοι και από τις πλατφόρμες που θα έχουμε, γιατί μπορούμε να κάνουμε πλατφόρμες ταξί χωρών, αλλά και με τρίτες χώρες, γιατί και τρίτες χώρες μπορούν να χρησιμοποιήσουν το ταμείο αυτό. Και ακριβώς γι' αυτό λέω πάντα ότι αυτό το ταμείο δεν είναι πατερναλιστικό, είναι μια σημαντική πρόκληση για την Ευρώπη και μια σημαντική πρόκληση και για άλλες χώρες. Μπορούν να γίνουν και διασυνοριακά προγράμματα. Μπορούμε να έχουμε πλατφόρμες θεματικές για αυτό το σκοπό. Όσον αφορά τις πληρωμές, πετύχαμε μια συμφωνία μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων για να έχουμε ένα σχέδιο πληρωμών, όπου το 2016 θα έχουμε 2 δισεκατομμύρια το πολύ απλήρωτα για το προηγούμενο δημοσιονομικό πλαίσιο. Στο τέλος αυτής της χρονιάς δηλαδή θα έχουμε 2 δισεκατομμύρια που θα είναι διαχειρίσιμο. Ξεκινάμε από την αρχή ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και κυρίως το Συμβούλιο θα τηρήσει τις υποχρεώσεις, πάκτα observanda, και μιλάμε για τη συμφωνία αυτή όσον αφορά τις πληρωμές. Όσον αφορά την διαδικασία επί του προπολογισμού. θα κάνω την ίδια προσπάθεια που έκανα και στις διαπραγματεύσεις. Και όπως είπα και στην αρχή, ο αγώνας συνεχίζεται. Αυτό τι σημαίνει. Αυτό σημαίνει ότι σε κάθε ε, διαδικασία του προπολογισμού θα προσπαθούμε να επανερχόμαστε στον στόχο, το έχω πει πάνω από 100 φορές, να ελαχιστοποιούμε τον αντίκτυπο πάνω στο Horizon 2020 και πάνω στο Connecting Europe. Μετά βέβαια πρέπει να δούμε ποιες είναι οι προτεραιότητες ποιο είναι το ποσό σε κάθε γραμμή, σε κάθε στόχο. Δεν μπορούμε τώρα να πούμε πόσα θα πάρουμε από το περιθώριο. Δεν γίνεται. Είμαστε ένα σκέλος της δημοσιονομικής αρχής και εμείς. Η άλλη αρχή είναι το Συμβούλιο. Αν ήμουνα μόνος μου, θα μπορούσα να δεσμευτώ με ένα νούμερο. Αλλά δεν είμαι μόνος μου. Πρέπει να υπάρξει συμφωνία με το Συμβούλιο για τον Προπολογισμό και για το 2016 το περιθώριο θα είναι περίπου ένα δις. ή λίγο παραπάνω. Αυτό είναι το συνολικό περιθώριο που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Θα συνεχίσουμε πάντως το έργο μας και το έργο μας είναι το ίδιο κάθε χρόνο. Σημειώνω πάντως ποια ποιες είναι δικές σας προτεραιότητες, ποιες είναι δικές σας προτάσεις. Και πιο συγκεκριμένα για τον στόχο μας αυτό και που τώρα θα επαναλαμβάνεται σε κάθε διαδικασία επί του προβλήσμου, κάθε χρόνο δηλαδή. Όσον αφορά τώρα τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς, έχω πει ότι δεν έχουν όλοι οι οργανισμοί τις ίδιες αρμοδιότητες ούτε και τις ίδιες ανάγκες. Άρα πρέπει να εξετάζουμε τον κάθε οργανισμό χωριστά. Αλλά υπάρχει κάτι που νομίζω ότι είναι ενδιαφέρον. Γνωρίζουμε πόσα μπορούμε να εξοικονομήσουμε όταν λέμε ότι θα κόψουμε τόσες θέσεις. Πρέπει όμως συγχρόνως να κοιτάμε πόσο θα κοστίσει αν κόβουμε αυτές τις θέσεις. Τι θέλω να σας πω, ότι μερικές φορές το να κόβουμε μια θέση κοστίζει πιο ακριβό από ότι αν δεν την κόψουμε αυτή τη θέση. Γιατί τι θα γίνει αν κοπεί αυτή η θέση, ποιες θα είναι οι επιπτώσεις. Το να μην κάνουμε κάτι μπορεί να έχει μια αρνητική συνέπεια πολύ αρνητική και άρα πρέπει να δούμε αυτή η αρνητική συνέπεια πόσο θα κόστιζε. Τουρισμός. Ε, φυσικά. Δεν υπάρχει γραμμή για τον τουρισμό. Είναι κάτι που καταλαβαίνω ότι είναι επίμαχο, αλλά σε αυτό τον προπολογισμό δεν έχουμε γραμμή για τον τουρισμό. Είναι εγκάρσιο. Τώρα για τα πειραματικά προγράμματα, τα πιλωτικά εξαρτάται από τα περιθώρια. Πάντως όλα τα πιλωτικά προγράμματα μπορούν να έχουν το πολύ 140 εκατομμύρια. Από όλες τις επιτροπές, ε, για όλες τις κατηγορίες, οι προπαρασκευαστικές δράσεις είναι 100 εκατομμύρια για τα πιλωτικά 140. Ε, Οπότε το σύνολο είναι 140. Πριν είχα πει ότι έχουμε ένα περιθώριο στην κατηγορία 1 που θα είναι λιγότερο από ό,τι τώρα, γιατί έχουμε τις επιπτώσεις του ΕΦΣΙ στο περιθώριο αυτό. Πρέπει να υπενθυμίσουμε και κάτι ακόμα, ότι στο στάδιο που βρισκόμαστε τώρα, έχουμε το σχέδιο προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πάνω σε αυτό συζητάμε, αλλά μετά το Συμβούλιο, και εδώ έρχομαι στη δημοσιονομική διαδικασία, το Συμβούλιο θα κάνει τη δικιά του ανάγνωση. Και μετά πάνω στην ανάγνωση του Συμβουλίου θα επιφέρουμε εμείς ε, τροποποίησεις, θα υποβάλουμε προτάσεις, τροποποίησεις, τροπολογίες. Και πρέπει να υπάρχει συνοχή. Γιατί το Συμβούλιο έχει εγκρίνει ένα δημοσιονομικό πολιετές πλαίσιο ομόφωνα. Και ομολογώ ότι μερικές φορές εκπλήσωμε γιατί χώρες οι οποίες έχουν εγκρίνει ένα πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο που προβλέπει κάθε χρόνο κάποια ποσά, το έχουν δεχτεί, γιατί ομόφωνα πάθηκε συμφωνία, μετά στη δημοσιονομική διαδικασία, ακόμα και με χαμηλότερο προπολογισμό εκφράζονται κατά. Και πολλές χρονιές χώρες μέλη είναι κατά του προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει συμβεί επανειλημμένα. Είναι μερικές χώρες που είναι πάντα κατά του προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακόμα και αν έχουν δεχτεί και εγκρίνει το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Εδώ λοιπόν θα ήθελα το Συμβούλιο να φέρεται με συνοχή απέναντι στις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει και το ίδιο να ισχύει και με τις δηλώσεις του. Για το Συμβούλιο κάνει πολλές δηλώσεις όπου μιλάει για την απασχόληση, για την νεολαία, για τη σύνδεση, για τις υποδομές και μετά δεν φροντίζει να βάλει επαρκή χρηματοδότηση. Θα δούμε. Έχουμε λοιπόν το σχέδιο προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τον Ιούλιο θα δούμε πού θα καταλήξει η ανάγνωση του Συμβουλίου, μετά έχουμε τη δικιά μας ανάγνωση και μετά θα προχωρήσουμε το χρονοδιάγραμμα όπως σας το είπα. Ότι δηλαδή αρχές Σεπτεμβρίου είναι προθεσμία για τις τροπολογίες στο κείμενο της Επιτροπής. Γιατί τώρα την εντολή θα ψηφίσουμε για τον τριμερή διάλογο. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα στις τροπολογίες επί του προπολογισμού. 3 Σεπτεμβρίου είναι προθεσμία. 23 Σεπτεμβρίου είναι για το ψήφισμα. 28, 29, 30 Σεπτεμβρίου θα ψηφίσουμε τον προπολογισμό για τις τροπολογίες. 12-13 Οκτωβρίου ψηφίζουμε το ψήφισμα και μετά στην Ολομέλεια 28 Οκτωβρίου και από τις 29 μέχρι την 1η Νοεμβρίου έχουμε τη συνδιαλλαγή για να καταλήξουμε σε κάποια συμφωνία. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς θα συνεχίσουμε το έργο μας, όχι μόνο γι' αυτό, για το χρονοδιάγραμμα, για τις τροπολογίες, τον προπολογισμό και για τις δικές σας προτεραιότητες, αλλά και μετά για τη συνδιαλλαγή, προκειμένου να καταφέρουμε να πετύχουμε αυτό στο οποίο όλοι αναφέρθηκαν, δηλαδή να επιστρέψουν στις γραμμές εκείνες που έχουν επηρεαστεί τα χρήματα τα οποία χρειαζόμαστε ώστε να τηρήσουμε και εμείς τις υποχρεώσεις μας βάσει του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Έτσι θα πετύχουμε τους στόχους μας που είναι στόχοι όλων μας. Το Connecting Europe είναι μια προτεραιότητα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Περιμένουμε τη συνέχεια. 13 και 14 Ιουλίου θα τοποθετηθούμε επί του σχεδίου αυτού έκθεσης και μετά θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή Μεταφορών. Ευχαριστώ. Περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Ανταλλαγή απόψεων για το ρουμανικό σιδηροδρομικό δίκτυο. Äh, Θα μας ενημερώσει για την κατάσταση των πραγμάτων στο σιδηροδρόμου της Ρουμανίας. Είχε παρετηθεί πρόσφατα ο, ο Ρουμάνος υπουργό Μεταφορών. Δεν είναι μαζί μας εδώ λοιπόν. Και γι' αυτό θα μας παρουσιάσει το θέμα ο εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Ρέτζιο. Κυρίες και κύριοι, Μαζί με τους συναδέλφους στην DG Move θα σας δώσουμε κάποιες συμπληρωματικές πληροφορίες για το Master Plan στις μεταφορές, το ρόλο που παίζει ε, στην Ευρώπη και τη σημασία που έχει το ρουμανικό Master Plan. Θα αναφερθώ σε τρία θέματα, τα οποία νομίζω ενδιαφέρον ιδιαίτερα και εσάς και κάποια από αυτά σας ανησυχούν θα έλεγα. Καταρχάς, τι είναι αυτό το Master Plan για τις μεταφορές. Ποιος είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ποια είναι η σχέση ανάμεσα στο Master Plan και στη χρηματοδότηση του νέου προϋπολογισμού στα πλαίσια ε, του ΕΣΥ Και ποιες είναι οι επιπτώσεις ανάμεσα σε αυτό και στον τομέα των σειροδρόμων, ιδιαίτερα στη Ρουμανία. Τι συνέπειες υπάρχουν σε σχέση με την χρηματοδότηση των σιδηροδρομικών προγραμμάτων στην Ρουμανία. Να πω πρώτα ότι το master plan αυτό, ξέρω ότι δεν είναι πρώτη φορά που ασχολείστε με το συγκεκριμένο θέμα και ξέρω ότι αρκετά μέλη έχουν συζητήσει το θέμα αυτό με την κυρία Κρέτου, την αρμόδια επίτροπο. Στην Επιτροπή είμαστε ικανοποιημένοι για τη συζήτηση αυτή και για την επίδειξη ενδιαφέροντος από πλευρά σας. Όσο, περισσότερη, θα έλεγα, όσο περισσότερο ενδιαφέρον δείχνετε, τόσο προσθέτεται στην νομιμοποίηση της παρουσίας μας στον διάλογο με τις ρωμανικές αρχές και με τις υπόλοιπες εθνικές αρχές. Ας περάσουμε τώρα σε ορισμένες βασικές αξίες, αρχές μάλλον. Στη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020 έχουμε μια σημαντική καινοτομία. Πριν αρχίσουμε δηλαδή εμείς να υιοθετούμε νέα προγράμματα, υπάρχουν ορισμένες προϋποθέσεις τις οποίες πρέπει να εκπληρούν τα κράτη-μέλη. Εμείς στο παρελθόν απλά υιοθετούσαμε τα προγράμματα, ενώ τώρα θα πρέπει να αποφασίσουμε αν ένα κράτος μέλος εκπληρεί ορισμένες προϋποθέσεις, είναι η λεγόμενη εκ των προτέρων ερεσιμότητα. Ε, μία από αυτές τις προϋποθέσεις είναι η ύπαρξη ενός πλαισίου μεταφορών. Ένα master plan για τις μεταφορές λοιπόν που καλύπτει το σύνολο των επενδύσεων μέχρι το 2030 σε όλα τα είδη των μεταφορών. Το ότι συνιστά σημαντική καινοτομία αποδεικνύεται από το ότι 20 χώρες έχουν αποφασίσει να επενδύσουν στις μεταφορές. Οι 18 από αυτές έχουν προς το παρόν συμμορφωθεί με τις προϋποθέσεις αυτές. Μόνο δύο, συγγνώμη, δύο. Η Σουηδία και η Κύπρος. We, uh, they themselves assessed with our help that they were και οι υπόλοιπε δεν έχουν συμμορφωθεί. Δηλαδή ή δεν έχουν ένα master plan ή έχουν κάποιο το οποίο δεν ήταν ε, συμβατό με τα επίπεδα τα οποία απαιτούνται. Θα ήθελα να πω ότι η διατύπωση του κανονισμού στο, στα πλαίσια των μεταφορών έχει συνταχθεί με ιδιαίτερη προσοχή από πλευράς του Συμβουλίου και των υπολείπων νομοθετών, ιδιαίτερα του Συμβουλίου. Είναι ένα στρατηγικό έγγραφο για το κράτος μέλος. Όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εμείς δηλαδή η Regio και η MOVE ε, έχουμε να παίξουμε και εμείς ένα σημαντικό ρόλο. Έχουμε προετοιμάσει κατευθυντήριες γραμμές. Ε, αν θέλετε, εμείς λέμε ποια είναι η μεθοδολογία που πρέπει να ακολουθηθεί. Υπάρχουν ορισμένα σετ κριτηρίων που πρέπει να γίνουν σεβαστά, όπως η δημόσια διαβούλευση, και οι προτεραιότητες ε, των επενδυτικών προγραμμάτων. Αν έχετε ερωτήσεις επιμέρους μπορώ να σας απαντήσω. Η Ρουμανία ήταν μία από τις χώρες οι οποίες ξεκίνησαν ενωρίς θα έλεγα πριν από την υιοθέτηση του κανονισμού ε, την επεξεργασία του Master Plan στον τομέα των μεταφορών. Ενεπλάκημεν και εμείς μαζί με άλλους ε, διεθνείς χρηματοδοτικούς μηχανισμούς όπως η Τράπεζα Επενδύσεων η Παγκόσμια Τράπεζα και μετά από πολλές ε, συζητήσεις και επαφές είμαστε σε μία φάση τώρα να διαπιστώσουμε ότι η Ρουμανία έχει προχωρήσει αρκετά. Είναι στην φάση της δημοσίας διαβούλευσης και θα πρέπει να καταλήξουμε στην τελική φάση στο τέλος του μήνα. Και μετά το επόμενο βήμα είναι να υιοθετηθεί σε πολιτικό επίπεδο από την Ρουμανική κυβέρνηση με κάποιον τρόπο. Είπα ήδη ότι πρόκειται για ένα εθνικό έγγραφο ουσιαστικά και εμείς μπορούμε να παρέμβουμε βέβαια και έχουμε παρέμβει μέχρι τώρα σε συμβουλευτικό επίπεδο εξηγώντας τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε. Υπάρχει κάτι όμως σε αυτό το master plan στο οποίο παίζουμε σημαντικό ρόλο ο εντοπισμός του καταλόγου των σημαντικών προγραμμάτων τα οποία θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος. Υιοθετούμε ένα πρόγραμμα για τις μεταφορές, εκεί όπου υπάρχει ένα μίξ προγραμμάτων και φυσικά έχουμε κάθε λόγο ε, να εντοπίσουμε και εμείς κάποιες προτεραιότητες και να είμαστε ιδιαίτερα δραστήριοι στον τομέα της ε, διευκρίνησης του ότι υπάρχουν δύο κριτήρια που παίζουν σημαντικό ρόλο για την κατάρτιση της λίστας των προτεραιοτήτων. Πρώτον, θα πρέπει να εντάσσεται στον πυρήνα των λεγόμενων TEN-T, των διευρωπαϊκών προγραμμάτων και δεύτερον να υπάρχει αυτό που ονομάζουμε οικονομική ε, ορατότητα, δηλαδή βιωσιμότητα και διαφάνεια. Έτσι λοιπόν πείσαμε τις ρωμανικές αρχές ότι αυτά είναι τα κριτήρια τα οποία θα πρέπει να γίνουν σεβαστά. Ένα σημείο το οποίο έχει δημιουργήσει κάποια ανησυχία στην Επιτροπή σας είναι οι επιπτώσεις που έχει το πρόγραμμα αυτό στους σιδηροδρόμους. Έχει υπάρξει στο εσωτερικό του Master Plan η ανάλυση της κατάστασης των σιδηροδρόμων της Ρωμανίας. Συμπέρασμα είναι ότι η μεταρρύθμιση του σιοδρομικού συστήματος είναι απαραίτητη. Are very in Romania. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο σιωδρομικό δίκτυο και δεν είναι βιώσιμη η διατήρηση όλων των γραμμών αυτών και είναι απαραίτητο να γίνουν ορισμένες στρατηγικές επιλογές Είμαστε σε διάλογο με τις ρωμανικές αρχές. Θεωρούμε ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία να υπάρξει μια περαιτέρω στρατηγική ανάλυση και μεταρρύθμιση του τομέα και πάντα εμείς λέμε ότι πριν ληφθεί η αδίποτε απόφαση για κλείσιμο ε, γραμμής, γιατί οι Ρωμάνοι θεωρούν ότι κάποιες γραμμές πρέπει να κλείσουν. Πριν ληφθεί η αδίποτε τέτοια απόφαση από την Ρουμανική κυβέρνηση απαιτείται μια πολύ προσεκτική ανάλυση για την οικονομική βιωσιμότητα του προγράμματος και για τις εκτιμήσεις του μεταφορικού έργου. Κάτι το οποίο θα ήθελα επίσης να υπογραμμίσω είναι ότι αυτό δεν επηρεάζει με κανένα τρόπο την σημασία και την συσχέτιση αν θέλετε ε, της στάθμισης, της χρηματοδότησης με τα συγκεκριμένα προγράμματα. Δηλαδή για την Ρουμανία ιδιαίτερα πιστεύουμε ότι πρέπει να διατηρηθεί το ίδιο ποσοστό χρηματοδότησης για τους σιδηροδρόμους με το ποσοστό που είχαμε το 2013. 38% της σύνολης χρηματοδότησης έχει σαν στόχο τα σιδηροδρομικά δίκτυα. και το ίδιο αυτό το 38% είναι το ποσοστό το οποίο προβλέπεται για την δημοσιονομική περίοδο την τρέχουσα, δηλαδή 14-20. Αν δείτε επίσης το Ταμείο Συνοχής, ένα από τα δύο ταμεία που εμπλέκονται, θα δείτε ότι το 50% του Ταμείου Συνοχής έχει σαν στόχο τους ιδεοδρόμους και το υπόλοιπο 50% οδικές και υπόλοιπες μεταφορές. Ιδιαίτερα τις ε, μεταφορές στο Δούναβι. Είναι λοιπόν αυτό ένα πολύ σημαντικό τμήμα του Ταμείου Συνοχής που στοχεύει, που τροφοδοτεί την, το μέσο Connecting Europe και ειδικά για τη Ρωμανία μετά φάσεις οι οποίες ελήφθησαν σήμερα αν δεν κάνω λάθος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα προγράμματα κατά προτεραιότητα 800 ε, εκατομμύρια δίδονται στην Ρουμανία για τους ιδεοδρόμους. Τα λέγω αυτά γιατί θέλω να επαναλάβω ότι είμαστε πλήρως αφοσιωμένοι στην εφαρμογή των κανόνων των ισιόντων έτσι ώστε να υπάρξει επαρκής χρηματοδότηση αυτού του είδους μεταφοράς που καθιστά για μας προτεραιότητα και δεν θα δεχθούμε η αδίποτε πρόταση μίασης της χρηματοδότηση του σιδηροδρόμου στη συγκεκριμένη χώρα. Και θα ευνοήσουμε, θα έλεγα, περαιτέρω μορφέ χρηματοδότηση. Ποια είναι τα επόμενα βήματα τώρα για την Ορμανία. Εμεί σύντομα θα υιοθετήσουμε το πρόγραμμα μεγάλων υποδομών, το οποίο περιλαμβάνει και την διάσταση τη μεταφορική, ε, είμαστε στην φάση των διαβουλεύσεων ανάμεσα στις διαφορετικές υπηρεσίες. Σε λίγες μέρες θα ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή και σχετικά με το Master Plan έχει προχωρήσει όπως σας είπα επαρκώς. Νομίζω ότι στο τέλος του 2015 θα ληφθούν όλα τα μέτρα έτσι ώστε η Ρουμανία να έχει το δικό της τελικό Master Plan. Αυτό το master plan δεν είναι ένα στατικό έγγραφο. Είναι μια στρατηγική η οποία βασίζεται σε ένα είδος αξιολόγησης του μεταφορικού έργου. Και όσο αλλάζει το μεταφορικό έργο θα αλλάζει φυσικά και το πρόγραμμα. Ο διάλογος θα συνεχιστεί, δεν τερματίζεται τίποτα στην παρούσα φάση είναι όμως ένα στρατηγικό έγγραφο το οποίο θα συνεχίσει να εξελίσσεται και με το οποίο εμείς εμπλεκόμεθα ε, επαρκώς. Θα μου επιτρέψετε να σταματήσω πλέον εδώ. Είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις και για τη Ρουμανία ή και γενικότερα για την κατάσταση των master plans και σε άλλες χώρες. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος, σας ευχαριστώ. Ο σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ που θέσατε αυτό το σημαντικό θέμα που νομίζω ότι όχι μόνο έφερε την Regio κοντύτερα στη Γενική Διεύθυνση MOVE αλλά και το αντίθετο και μια συνεργασία δηλαδή μέσα από τις διαρκείς συζητήσεις που διεξάγουμε με τις ρουμανικές αρχές για την υλοποίηση του master plan. Τα αποτελέσματα είναι θετικά δεν έχουν ακόμα λάβει οριστική μορφή, αλλά έχουν ήδη υποβληθεί σε πολλούς από εμά και σε σημαντικούς stakeholder. Λίγα λόγια για τον παραλληλισμό με την πραγματική πολιτική. Στο σύνολό της η Ρουμανία αποτελεί ένα στέρεο εταίρο σε ό,τι αφορά την πολιτική του σιδηροδρόμου. Και στο Master Plan φάνηκε από απόλυτα ε, σταθερή στην υλοποίηση των προγραμμάτων TNT έχει παίξει το ρόλο της για την υλοποίηση των σχεδίων των διαδρόμων, των δύο διαδρόμων δηλαδή που διέρχονται την χώρα έχει κατανοήσει επίσης απολύτως τις προτεραιότητες που θέλαμε, θέλησαμε δηλαδή ε, να τις υποβάλουμε και όπως είπε η συνάδελφός μου στη συζήτηση που θα κάνετε την επομένη Δευτέρα το βράδυ νομίζω στο Στρασβούργο με τον Επίτροπο Μπούλς τα αποτελέσματα των εργασιών μας με τη Ρουμανία είναι πολύ τα θετικά. Η Ρουμανία στην πρώτη φάση χρησιμοποιεί 70% της χρηματοδότησης από τον εθνικό φάκελο και τα περισσότερα από τα έργα είναι πραγματικά έργα και πολύ σημαντικά έργα ε, διαμεθοριακών σιδηροδρομικών διασυνδέσεων που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν, ελείπουν. Το άλλο, η άλλη πτυχή είναι η, πολιτική της, είναι η πτυχή της πολιτικής. Η Ρουμανία ήταν πάντοτε μέρος και του τεχνικού πυλώνα αλλά και του πολιτικού πυλώνα της ε, πολιτικής σιδηροδρόμων στο σύνολό της και ως κυβέρνηση και ως δημόσιος τομέας. Τέλος, για την αναδιατύπωση Μόνο τρεις χώρες μέλη έχουν έτσι και λίγο κυρώσει και μεταφέρει μέχρι τώρα τον, την αναδιατύπωση του κανονισμού, όμως εφαρμόζει το περιεχόμενό του έτσι ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση στη χώρα με σημαντικές μεταρρυθμίσεις που έχουν ήδη αρχίσει και συνεχίζονται. Δύο παραδείγματα. Το πρώτο είναι η, η πλήρης λογική των μάνατζερ της υποδομής, δεν κλείνουν δηλαδή οι οι γραμμές μόνο και μόνο για να τις κλείσουν, αλλά προβλέπεται η υποχρέωση, εφόσον κλείνουν κάποιες γραμμές, αυτό να γίνεται σύμφωνα με μία σε βάθος ανάλυση της κατάστασης και από οικονομική δημοσιονομική σκοπιά και από άποψη ε, μεταφορών. Δεύτερο, το master plan της Ρουμανίας προτείνει σε βάθος επανεξέταση της ε, κατάστασης των δημόσιων μεταφορών της και με ειδικό οργανισμό στα πλαίσια του ρωμαϊκού Δημοσίου που θα έχει μάλιστα και ισχυρές εξουσίες για να μπορέσει να επιτύχει την επανεξέταση αυτή μέσα σε μια χώρα η οποία έχει ισχυρά σιδηροδρομική παράδοση, ενώ τη Ρουμανία φυσικά, και έχει παραγάγει και διάφορες ε, σχετικές δραστηριότητες και ε, να αντιμετωπιστούν πραγματικά οι ανάγκες του κόσμου, του κοινού. Μάλιστα, λέει ο κ. Κράμερ, ορισμένοι έχουν ζητήσει ήδη το λόγο. Επισημαίνω μόνο ότι είχαμε ομόφωνα συναποφασίσει να κάνουμε τη σε αυτή μαζί με τη συνάντηση των συντονιστών και μετά απευθύναμε επιστολή στην Επίτροπο και λάβαμε απάντηση που δεν είναι ικανοποιητική όμως γιατί μας λέει ότι δεν πρόκειται να μας αποσταλούν τα έγγραφα. Έχουμε όμως εμείς το δικαίωμα ως κοινοβουλευτική επιτροπή του Κοινοβουλίου να ε, δούμε τα έγγραφα Όμως στην, επιστολή, στην απαντητική επιστολή μας λέει ότι αυτά συζητούνται ακόμα με τη ρουμανική κυβέρνηση. Έχουμε όμως από τη συνθήκη το δικαίωμα να εξετάσουμε τα έγγραφα. Δεν μπορείτε να πείτε ότι αυτά τα έγγραφα δεν μπορείτε να τα δείτε, είναι δικαίωμά μας και το δικαίωμά μας αυτό το διεκδικούμε. Έχετε και την επιστολή μας, την βλέπετε και τώρα ναι, ο Μάριαν. Ευχαριστώ αγαπητέ Πρόεδρε. Γνωρίζω ότι το βασικό θέμα της συζήτησης είναι ο σιδηρόδρομος μέσα από το master plan. Αλλά έχω και μια ερώτηση για το νοοδικό χάρτη του master plan και που συνδέεται με τα όσα είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν. Είπε δηλαδή ότι τα δυο κριτήρια που έλαβαν υπόψη το, το βασικό δίκτυο και η οικονομική βιωσιμότητα. Αυτό που θα πρέπει να εγκριθεί στο μεγάλο επιχειρησιακό πρόγραμμα υποδομών για τους δρόμους στη Ρουμανία περιλαμβάνει τουλάχιστον 12 έργα από τα οποία τα 5 είναι βασικό δίκτυο, δίκτυο πύρινας τα υπόλοιπα είναι εκτός. Και αυτό δεν συμβαδίζει με τα κριτήρια που μας είπαν εδώ. Κάτι άλλο τώρα. Θέλω να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει την εναρμόνιση του ρουμανικού master plan με τους γείτονές της, με τους γείτονές της χώρας. Ώστε να μην έχουμε από τη μια μεριά των συνόρων ας πούμε ένα αυτοκινητόδρομο και από την άλλη μεριά τίποτα. Μέχρι το 2030 για τη Ρουμανία. Η Κομισιόν λέει ότι το master plan είναι ευθύνη των χωρών μελών. Ταυτόχρονα όμως εγκρίνει κατάλογο έργων προτεραιότητας. Ο κατάλογος έργων προτεραιότητας στο μεγάλο επιχειρησιακό πρόγραμμα για τις μεταφορές, για τις υποδομές δηλαδή. Αυτό σημαίνει ωστόσο ότι είναι ευθύνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να εγκρίνει τις, παρα... προτεραιότητες του κανονισμού TEN-T, των ευρωπαϊκών δικτύων δηλαδή. Γι' αυτό θέλω να μάθω ποια θα είναι η απόφαση για το οδικό master plan στη Ρουμανία και αν πρόκειται να πληρώσουν τα κριτήρια τα οποία ήδη έχουν ανακοινώσει. Ο πρόεδρος Κράμερ. Δεν συζητούμε όμως τώρα το Road Master Plan, το Master Plan για τους δρόμους. Έχουμε ζητήσει να προσέλθουν τα πρόσωπα αυτά εδώ για να μιλήσουμε για το σιδηροδρομικό δίκτυο. Γιατί ακούσαμε ότι πρόκειται να κλείσουν το 40% του σιδηροδρομικού δικτύου. Αυτό είναι το συγκεκριμένο ε, ζήτημα τώρα και όχι συνολικά οι καταστάσεις μεταφορών στη Ρουμανία τα Ταπαντέλ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ξεκινήσω ευχαριστώντας την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για τις πληροφορίες που μας έδωσε και για τη συνεργασία ανάμεσα στις Ρωμανικές Αρχές και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα να κάνω κάποιες παραπομπές θα έλεγα στη συγκεκριμένη έκθεση σχετικά με τα ειδικά χαρακτηριστικά του ρουμανικού σιδηροδρόμου. 11.000 ε, χιλιόμετρα. Είναι το 7ο δίκτυο σε μήκος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα τμήμα ανήκει στα δίκτυα TEN-T και ανάμεσα στο 2010 με το 2015 το δίκτυο ε, μειώθηκε κατά 5% ενώ το ευρωπαϊκό δίκτυο κατά 7,8% λιγότερο από άλλες μειώσεις άλλων χωρών που δεν θα τις αναφέρω τώρα αλλά τη βρίσκεται στη σελίδα 7. Νομίζω λοιπόν ότι μία συζήτηση ε, θα πρέπει να διευρύνει το αντικείμενό της και να συμπεριλάβει τον τρόπο με τον οποίο οι σιδηροδρομικές υποδομές μειώνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εμείς θέλουμε αηφορία στις μεταφορές. Η αηφορία έχει σαν βασικό στόχο τη μείωση των εκπομπών και θα πρέπει αυτό να αφορά το σύνολο της Ένωσης και όχι μόνο την Ρωμανία. Μιας και βρισκόμαστε λοιπόν στην κατάσταση αυτή, να σας πω ότι το Master Plan παίζει σημαντικό ρόλο για τις μεταφορές στη χώρα αυτή και οι προτεραιότητες περιλαμβάνονται και γίνονται δεκτές σαν βάση για τη χρηματοδότηση από πλευράς Ένωσης. Το έγγραφο αυτό έχει σαν στόχο την βελτίωση της αηφορίας του δικτύου, την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών, και την ενθάρρυνση καλύτερης λειτουργίας των ε, επιχειρήσεων που διαχειρίζονται το δίκτυο. Το δίκτυο αυτό δεν θα πρέπει να αντιμετωπιστεί σαν ένα δίκτυο προς απομείωση, αλλά θα πρέπει ε, να εξελιχθεί και να αναπτυχθεί. Φυσικά και απαιτούνται μεταρρυθμίσεις, όπως το είπαν άλλωστε και οι εκπρόσωποι της Επιτροπής, έτσι ώστε τα δίκτυα τα οποία είναι διαθέσιμα να μπορέσουν να λειτουργήσουν με καλύτερους και ποιοτικότερους όρους παρέχοντας καλύτερες υπηρεσίες. Αυτό προϋποθέτει την εκ των προτέρων ερεσιμότητα της ανάπτυξης του δικείου. Χωρίς αυτή τη χρηματοδότηση το δίκτυο το ρουμανικό δεν θα μπορέσει να εξυπηρετήσει καλύτερα και περισσότερους επιβάτες. Οι στόχοι τώρα για τις εκπομπές και είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει χωρίς την έγκριση του Master Plan έτσι ώστε να καλύψουμε τις ανάγκες του συνόλου των τρόπων μεταφοράς μεταξύ των οποίων του σιδηροδρομικού δικτύου. Καλό θα ήταν λοιπόν να συγκεντρώσει κανείς την προσοχή του στο τελικό στόχο έτσι ώστε μια πολιτική ε, όπως αυτή της Ρουμανίας να βοηθήσει να βελτιώσει την κατάσταση ενός τομέα σημαντικού αλλά αναποτελεσματικού και να γίνει αποτελεσματικός, αηφόρος και ασφαλής. Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις, ε, όχι πολύ ενθαρρυντικές και από τις άλλες χώρες και γι' αυτό θα πρέπει να δούμε τι ανάγκες μπορούμε να καλύψουμε σε επίπεδο χρηματοδότησης. Να επαναλάβω αυτά τα οποία έχω πει, ότι στην παρούσα φάση έχουμε μία ανάγκη ανάπτυξης των υποδομών για το σύνολο των ειδών μεταφορών, ιδιαίτερα για τις χώρες οι οποίες βρίσκονται στα άκρα της Ένωσης και οι οποίες έχουν ανάγκη από περισσότερη ενέργεια για την ανάπτυξη των δικτύων τους. Ερτογκ. Äh, Ευχαριστώ πρώτα για την ενημέρωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, των δύο Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συντονιστής εγώ και έχω παρακολουθήσει από την αρχή τη συζήτηση αυτή. Αν ήμουν δημοσιογράφος θα έλεγα τώρα θα έλεγα προς Θεού κάνετε λάθος. Διότι κάποιοι εδώ προσπαθούν να ξεμπροστιάσουν μια χώρα. Οι τοποθετήσεις των εκπροσώπων της Κομισιόν δείχνουν ότι όντως δεν συμβαίνει αυτό. Τα έφυγε η κυρία Ταπαντέλ. Ως Ευρωπαίος πολιτικός θα ήθελα τα πράγματα να είναι διαφορετικά. Ωστόσο, εξακολουθεί ο σχεδιασμός των μεταφορών να είναι εθνική πολιτική. Μήπως εμείς θα τολμούσαμε να πάμε να υπαγορεύσουμε στους Γερμανούς τι θα κάνουν στην πολιτική μεταφορών τους το ίδιο πρέπει να ισχύει και για οποιαδήποτε άλλη χώρα και για τη Ρουμανία. Πού ήταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή Μεταφορών όταν το 1994 στη Γερμανία μειώθηκε μαζικά το σιδεοδομικό δίκτυο. Σήμερα τα επικρίνουμε αυτά που έγιναν τότε. Τότε δεν είχαν πει, δεν είχαν μιλήσει πολύ. Θέλω λοιπόν αυτά να ληφθούν υπόψη και τέτοια λαϊκι, τέτοιοι λαϊκισμοί να μην έχουν ε, τόπο εδώ. Ο πρόεδρος. Κοιτάξτε, μια πολιτική ομάδα ομάδων πράσινων ζήτησε να συζητηθεί το θέμα. Γράψαμε γράμμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ζητήσαμε πληροφορίες. Και πληροφορίες δεν λάβαμε, παρόλο που ε, είναι δικαίωμά μας. Μάθαμε ότι πρόκειται να κλείσουν το 40% του σιδηροδομικού δικτύου. Θέλαμε επιβεβαίωση μα είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δεν έχει ιδέα και ότι αυτό είναι καθαρά θέμα των Ρουμάνων. Από την άλλη μεριά ακούγαμε πληροφορίες ότι αυτό το κλείσιμο το έχουν συζητήσει και συμφωνήσει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και θέλαμε λοιπόν να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Αυτό ήταν το αίτημά μας. Το αίτημά μα αυτό το στήριξαν στην συνάντηση συντονιστών όλοι οι συντονιστέ. Και εσείς κύριε Ερτούκ, συντονιστή των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Καλύτερα να έχει γίνει βέβαια μία εβδομάδα πριν να ληφθεί η επιστολή. Αλλά και τα έγγραφα. Και τα είχαμε συζητήσει όλα αυτά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτοί λένε ότι είναι καθαρά από των Ρουμάνων. Αλλά αυτό δεν είναι σωστό. Εμείς ως Ευρωβουλευτές έχουμε και το δικαίωμα και το καθήκον να βρούμε την αλήθεια. Γι' αυτό διεξάγεται η σημερινή συζήτηση. Αν τώρα η συζήτηση αυτή είναι λαϊκιστική, κοιτάξτε, ο καθένα μπορεί να έχει τη γνώμη του και είναι ελεύθερο. Αυτό που θέλουμε εμεί πρώτα-πρώτα είναι τα γεγονότα. Συγκεκριμένα γεγονότα μπορώ να τα κρίνω κι εγώ. σε αυτό το κλείσιμο σιδηροδρομικών γραμμών δεν υπάρχει καμία γραμμή που να έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αμφιβάλλω πολύ ότι είναι έτσι, διότι η Ρουμανία για τους ιδιοδρόμους έχει λάβει συγχρηματοδότηση 85% από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν λοιπόν έχει δοθεί χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 85% δεν, μπορεί, δεν είναι καθαρά ρουμανικό θέμα. Γι' αυτό ρωτώ ποιες διαδρομές έχουν κλείσει, γιατί στην επιστολή σας λέτε τα μεγαλύτερα έργα και όχι όλα, μπορείτε να μου διασφαλίσετε ότι καμία γραμμή δεν θα κλείσει από αυτές που έχουν συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν πάμε να χρηματοδοτήσουμε, να συγχρηματοδοτήσουμε υποδομές οι οποίε μετά θα κλείσουν. Αυτές οι ερωτήσει είναι σημαντικές. Εδώ στο φυλάδιο αυτό, ορίστε, που έχει μέσα και σχέδιο των σιδηροδρομικών γραμμών της Ρωμανίας, έχει εδώ και μια σημαντική γέφυρα ανάμεσα στην Ουγγαρία και στη Ρουμανία παρόλο που για πολλές δεκαετίες ήταν σοσιαλιστικά αδέρφια, μία μόνο γέφυρα υφίστατο. Τώρα με χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης φτιάχτηκε άλλη γέφυρα, που δεν τη βλέπω εδώ, γέφυρα η οποία είναι και για αυτοκίνητα και για σιδηροδρόμους. Είναι εθνικό θέμα αυτό ή είναι θέμα διασύνδεσης δυο χωρών μελών που έχει το στόχο να τις προσεγγίσει περισσότερο. Αυτό είναι σημαντικό και ιδίω για τα έγγραφα. Δεν επιτρέπεται, δεν μπορούμε να δεχτούμε κάτι τέτοιο. Έχουμε το δικαίωμα ως ευρωβουλευτέ να εξετάσουμε τα έγγραφα. Αν τώρα θα τα χαρακτηρίσουν εμπιστευτικά είναι μια άλλη υπόθεση. Δεν μπορούν να πούν απλώ α, πρόκειται για αλληλογραφία μεταξύ Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Ρουμανία, διότι αυτή η τελική παράγραφο του εγγράφου είναι παραπλανητική. Διότι και οι πολίτε έχουν βεβαίω δικαίωμα να ελέγχουν τα έγγραφα, αλλά όχι όπω οι βουλευτέ. Οι βουλευτέ καταρχήν Τώρα κοιτάξτε, εσείς κύριε Τούκπαλη, αναγκάζομαι να λάβω το λόγο γιατί δύο φορές αναφερθήκατε στο όνομά μου. Τη μορφή του λαϊκισμού δεν θα απαλλαγείτε από αυτήν εσείς οι πράσινοι, διότι σωστά είναι τα ερωτήματα που θέτετε. Τώρα τα λέτε όμως. Εάν η διαδικασία έχει κινηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να έχουν γίνει ερωτήσεις πριν, τότε θα μας ενδιαφέρει πράγματι η ουσία γιατί όπως έγινε όμως το πράγμα από την αρχή ήταν καθαρά λαϊκιστικό παιχνίδι για να απευθυνθεί μομφή σε μια κυβέρνηση μιας χώρας μέλους. Εγώ είπα από την αρχή ότι η διαδικασία δεν έχει καλώς και η διαδικασία δεν θα πρέπει να προχωρήσει, κατά αυτόν τον τρόπο. Η τύχη στην πλειοψηφία των συντονιστών. Αυτό είναι απολύτως καθαρό εξακολουθώ να επιμένω ότι πρόκειται για λαϊκισμό. Ο πρώτο Κράμερ. Δεν είναι ακριβώς τα πράγματα έτσι. Εμείς ζητήσαμε πληροφορίες και ζητήσαμε και προτίσαμε να τι λάβουμε. Και επειδή δεν τις λαμβάναμε, γι' αυτό στην συνάντηση των συντονιστών αποφασίσαμε να γίνει η παρούσα συνεδρίαση. Ήταν ομόφωνη η συνεδρίαση. Μετά προέκυψε η ένσταση. Όχι όταν είπαμε ότι θα λάβουμε την απόφαση για να ζητήσουμε και να λάβουμε τις πληροφορίες τις οποίες είχαμε ήδη ζητήσει γραφτός. Αυτά περί λαϊκισμού ο καθένας σας τα βλέπει όπως θέλει. Εμένα με ενδιαφέρει η ουσία. Ένα πράγμα είναι ξεκάθαρο. Όταν κλείνουμε μια σιδηροδρομική γραμμή, εγώ δεν ξέρω κανένα αυτοκινητόδρομο που να έχει κλείσει στη Ρουμανία ή στη Βουλγαρία, πάντα το ψαλίδι πέφτει στον, στον σιδηρόδρομο. Και όμως οι μεταφορές προσώπων είναι τη τάξη του 72% στον σιδηρόδρομο. Η Κλάουδια τα τι πάρει το λόγο. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι είναι απόλυτα φυσιολογικό να τα συζητάμε αυτά τα θέματα, αλλά οι σιδηρόδρομοι φτιάχτηκαν με ευρωπαϊκά χρήματα. Τα χρειαζόμαστε τα ευρωπαϊκά χρήματα για να συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε τις δρομικές ε, υποδομές και να τις συντηρούμε δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό, πρέπει να το γνωρίζουμε. Υπάρχει μεγάλη διαφορά εδώ και ένα μεγάλο σφάλμα που κάνουμε. Χρειαζόμαστε χρηματοδότηση για να αναπτύξουμε τις υποδομές στο σύνολό τους, είτε σιδηροδρομικές ή άλλων ειδών μεταφοράς. Δεν θέλουμε να κλείσουμε τη ροή αυτή χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα έχει τη δυνατότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαντήσει και αναμένουμε μεγάλο ενδιαφέρον τι θα πει. Να διευκρινίσω τα ορισμένα πράγματα. για τους σιδηροδρόμους που χρηματοδοτήθηκαν και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση να κλείσουν υποδομές τις οποίες έχουμε συγχρηματοδοτήσει, σας το λέω αυτό επισήμως. Σιδηρόδρομοι που έχουν συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα διατηρηθούν. Έχουμε μάλιστα και την δέσμευση της Ρουμανικής κυβερνήσεως ότι ένα ποσοστό του ΑΕΠ θα διατίθεται ετησίως για την διατήρηση, για τη συντήρηση δηλαδή των σιδηροδρομικών αυτών γραμμών. Σε αυτό είμαι σαφέστατη. Μιλήσατε ακόμη ρωτήσατε μάλλον, ποιος είναι ακριβώς ο ρόλος της Κομισιόν. Εμπλέκεται η Κομισιόν ή όχι στο Master Plan. Θα προσπαθήσω να διευκρινίσω. Το Transport Master Plan είναι στρατηγικό, εθνικό στρατηγικό έγγραφο. Αυτό που κάνουμε εμείς της Κομισιόν είναι ότι παρεμβαίνουμε για να δούμε, για να καθορίσουμε εάν υπάρχει ή όχι συμμόρφωση με ορισμένες προϋποθέσεις. Υπάρχουν κάποια κεντρικά κριτήρια και μια μεθοδολογία ότι δηλαδή το Transport Master Plan θα πρέπει να συμμορφώνεται με αυτά τα κριτήρια. Δεν παρεμβαίνουμε στις εθνικές επιλογές. Έχουμε λόγο όμως σε θέματα μεθοδολογίας και εφαρμοζομένων κριτηρίων. Παράδειγμα, αν μια χώρα μέλος μας υποβάλλει ένα Transport Master Plan το οποίο δεν έχει συζητηθεί καθόλου στη χώρα μέλος, εμείς τότε θα προβάλλουμε ένσταση, διότι μια στρατηγική δεν μπορεί να είναι απλά η στρατηγική ενός μεμονωμένου υπουργού, θα πρέπει να είναι της κυβέρνησης της χώρας. Για παράδειγμα, το κριτήριο της δημοσίας συζητήσεως και του τι προκύπτει από μια δημόσια συζήτηση είναι ένα κρίσιμο κριτήριο. Άλλωστε, μεταξύ άλλων, Εάν ένα transport master plan βασίζεται μονάχα σε νούμερα και όχι σε ένα μοντέλο συγκοινωνιών, πάλι εκεί παραβιάζεται ένα κριτήριο. Λέμε λοιπόν, είναι εθνικό στρατηγικό σχέδιο, αλλά πρέπει να συνταχθεί με ορισμένε παραμέτρους, κάτω από ορισμένε προποθέσει. Να έρθω σε ένα άλλο θέμα που σας απασχολεί την αίτηση προς τους επιτρόπους Κρέτσο και Μπούλς για πρόσβαση σε έγγραφα. Όσον αφορά τα ίδια τα Transport Master Plan, τα έγγραφα αυτά είναι διαθέσιμα στο κοινό. Και σας έχουμε δώσει την ιστοσελίδα ειδικώς για τη Ρουμανία. Γενικώ όμως υπάρχουν. Αν σας, ενδιαφέρουν περισσότερα πράγματα, σας ενδιαφέρει η αλληλογραφία. Αυτό που προσπάθησε να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι να συμπεριλάβει την ουσία της αλληλογραφίας στο έγγραφο. Είπαμε μετά, επειδή ακόμη βρισκόμαστε εσωτερικά μέσα στη διαδικασία λήψης αποφάσεως πάνω σε ένα πρόγραμμα, μιλούμε δηλαδή εδώ για την απόφαση της Κομισιόν επί του προγράμματος έγκρισης της λίστας των έργων. Θεωρήσαμε λοιπόν ότι επί του παρόντος πλήρης πρόσβαση σε αυτή την αλληλογραφία δεν μπορεί να δοθεί διότι θα παρέμβει με τον τρόπο αυτό στην διαδικασία λήψης των αποφάσεων. Όταν θα εγκριθεί βέβαια το πρόγραμμα τότε αλλάζει η ανάλυση και θα επανέλθουμε στους επιτρόπους Κρέτσου και Μπούλς να δούμε σε λίγες μέρες τι μπορεί να γίνει έτσι ώστε να σας δώσουμε πρόσβαση στα έγγραφα. Και βεβαίως είμαστε δεσμευμένες και εμείς για πλήρη διαφάνεια, ιδίω απέναντι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα εξετάσουμε λοιπόν την κατάσταση όταν θα έχει εγκριθεί το πρόγραμμα. Για τις άλλες παρεμβάσεις νομίζω ότι αποτελούσαν μάλλον σχόλια. Δεν θα τοποθετηθώ λοιπόν. Είναι σημαντικό, όπως είπαμε, να εξετάσουμε όχι μοναχά το ρουμανικό master plan και τις μεταρρυθμίσεις, αλλά όλα τα master plan της περιοχής. Και ένα σημαντικό πράγμα είναι ότι ενθαρρύνουμε και ακόμη περισσότερο από ενθαρρύνουμε τις όμορες χώρες μέλη να προβαίνουν σε διάλογο. Διότι αν θέλουμε να δημιουργηθούν οι διάδρομοι, βεβαίω πρέπει να συνομιλούν οι όμορες χώρες μέλη. Γι' αυτό χρειάζονται όμως τα master plan για τις μεταφορές για να εξασφαλίσουμε ότι θα ολοκληρωθούν και όλες οι διάδρομοι. Που είναι και σημαντικό μέρος της ε, διευκόλυνσης συνδέοντας την Ευρώπη. Αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ ο κύριος Ονίλη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δύο λόγια ακόμα. Πρώτον, όπως υπογράμμισα και στην εισαγωγή μου, το ότι τέθηκε το θέμα ήταν χρήσιμο. Δεν έχουμε την ε, εξουσία να εγκρίνουμε εμεί το master plan για, αντί για μία χώρα μέλος, έχουμε όμως ε, την δυνατότητα να επηρεάσουμε. Και νομίζω ότι χάρη στα όσα επιπλέον υπογραμμίσαμε για το θέμα, έχουμε μπορέσει να βελτιώσουμε την ποιότητα του master plan. Είμαστε ευγνώμονες στις ρουμανικές αρχές για τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετώπισαν το θέμα καθόλου το εγχείρημα, αλλά και για τα αποτελέσματα, γιατί όπως είπα το master plan ευθυγραμμίζεται πλήρως με τα διευρωπαϊκά δίκτυα, τουλάχιστον από τη δικιά μας την πλευρά, και αναφέρεται στον πρώτο κατάλογο προτεραιοτήτων που έχει υποβληθεί. Ο κατάλογος των προγραμμάτων είναι στη διάθεσή σας από σήμερα το πρωί, πρέπει να ξέρετε. Το έχουμε στείλει επίσημα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα σχέδια προγραμμάτων που σκοπεύουμε να στηρίξουμε οικονομικά, δηλαδή βάσει των συζητήσεων που θα έχετε και εσείς με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την επόμενη εβδομάδα. Αυτή η πληροφορία δηλαδή είναι στη διάθεσή σας. Επίσης, η απειλή του να κλείσει 40% του δρομικού δικτύου σε αυτήν την τόσο σημαντική χώρα σιδηροδρομικά ήταν κάτι βέβαια που μας ανησύχησε. Με το Master Plan υπάρχει δυνατότητα να κλείσουν κάποιες γραμμές, αλλά δεν έχουν αποφασιστεί σε αυτό το στάδιο, ε, δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις για να κλείσουν γραμμές. Αν γίνει αυτό, θα είναι σύμφωνα με την συνολική νομοθεσία και η υποχρέωση θα υπάρχει για τον διαχειριστή να αποδείξει ότι δεν υπάρχει οικονομικό όφελος από αυτές τις διάφορες διαδρομές. Επιπλέον, το κλείσιμο έχει να κάνει με πρόβλημα χρηματοδότησης για τη συντήρηση. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, δεν έχουμε τόσα πολλά μέσα για να μπορούμε να βοηθήσουμε οποιαδήποτε χώρα να συντηρήσει την υποδομή της. Έχουμε όμως άλλα μέσα, τα οποία με τη Γενική Διεύθυνση Ρέτζιο θα χρησιμοποιήσουμε για να βοηθήσουμε τη χώρα να χρησιμοποιήσει όσο γίνεται καλύτερα το δίκτυο όσο έχει σήμερα και να φροντίσουμε να αναπτυχθεί περισσότερο προς το συμφέρον όλων των ε, χρηστών. Είτε πρόκειται για τους επιβάτες, είτε πρόκειται για όσους ε, μετακινούν εμπορεύματα. Ευχαριστώ. Πού είναι το έγγραφο, ποιο είναι το έγγραφο που λέτε ότι λάβαμε σήμερα το πρωί. Εγώ γνωρίζω μόνο την επιστολή που περιλαμβάνει λίστα των πιο σημαντικών έργων. Αλλά μόνο αυτό, δεν έχουμε πλήρη κατάλογο. Πότε έλθε σήμερα το πρωί. Σας διαβάστη σήμερα το πρωί. Λόγω του δικαίωματός σας κοινοβουλευτικού ελέγχου και για τις συζητήσεις που θα διεξαγάγετε με τον Επίτροπο την Δευτέρα και για την Επιτροπή ΣΕΦ για να έχετε χρόνο να εξετάσετε τον κατάλογο των έργων που προτείνουμε να χρηματοδοτηθούν και να έχετε και τη δυνατότητα να απαντήσετε να έχετε τη δυνατότητα να θέσετε ερωτήσεις και να σας απαντήσουμε εμείς. Κράμερ. Ωραία. Εδώ λίγη συζήτηση αυτή. Τώρα. Το επόμενο θέμα. Το υπαριθμό 6 follow-up στην πτώση του αεροσκάφους της German Wings με εκπροσώπους της ΕΑΖΑ, Κομισιόν. Πάτε εκεί, παρακαλώ ελάτε εδώ. Ich begrüße sehr herzlich Herrn Philipp Cornelius. Καλώς ήρθατε κύριε Φίλιπ Κορνέλιους, τη για την ασφάλεια πτήσεων στη DigiMove, καθώς και τον εκτελεστικό διευθυντή της ΕΑΣΑ. Ποιος επιθυμεί να, να αρχίσει, συγγνώμη. Πάτε εκεί, όχι εσείς. Α, ο κύριος Κορνέλιους. Αγαπητά μέλη, μετά από την πτώση της πτήσης της German Wing τον Μάρτιο που κόστησε στη ζωή σε 150 περίπου άτομα, οι σκέψεις μας πηγαίνουν στις οικογένειες των θυμάτων. Ήταν ένα πάρα πολύ σπάνιο συμβάν στην ιστορία των αερομεταφορών και ένα ιδιαίτερα τραγικό συμβάν. Μετά από τρεις μήνες που βρισκόμαστε, η προκαταρκτική έκθεση από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Γαλλίας λέγει ότι η πτώση τη συγκεκριμένου αεροσκάφους προκλήθηκε από σκόπιμη ενέργεια του συγκυβερνήτη. Να προσθέσω ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία έρευνας και αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Ότι δηλαδή θα πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία και θα λάβουμε τότε υπόψη τις συστάσεις τις οποίες θα εκδώσει η Γαλλική ερευνητική αρχή. Γνωρίζετε ότι ανακοινώθηκε από, την, από δικαστικές πηγές ότι γίνεται και σε επίπεδο νομικό, δικαστικό, μια έρευνα ανάκριση η οποία εξετάζει τα πρόσωπα και τις επιχειρήσεις στη Γαλλία ή ουδήποτε αλλού ε, μπορεί να είναι υπεύθυνε για το ατύχημα αυτό. Ε, η Επιτροπή δεν εμπλέκεται βέβαια άμεσα, αλλά παρακολουθούμε όμως τα θέματα της έρευνας στον τομέα της ασφάλειας. Είναι βασικό για μας για να κατανοήσουμε τις αιτίε και τους παράγοντες που συνεισφέρουν ε, στο ατύχημα. Η σκόπιμη δράση λοιπόν του συγκυβερνήτη έφερε στην επιφάνεια τα θέματα της ιατρικής καταλληλότητας, της ιατρικής κατάστασης και της πρόσβασης δεύτερο θέμα στο, στο ε, τμήμα του αεροσκάφους που βρίσκεται ο κυβερνήτης και ο συγκυβερνήτης. Επίτροπος Μπούλτς ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας των Αερομεταφορών να εξετάσει τα δύο θέματα αυτά, δηλαδή το κλείδωμα της πόρτας του κόκπιτ και τα κριτήρια και τις διαδικασίες για την ιατρική παρακολούθηση της καταλληλότητας της σωματικής ε, των κυβερνητών. Η διαδικασία αυτή συνεχίζεται, συμμετέχουν εκπρόσωποι των αρχών ε, για, την αερομε... για τις αερομεταφορές από διάφορες χώρες και ο κύριος θα αναφερθεί σε αυτά πιο αναλυτικά. Η προσπάθεια της Task Force γίνεται παράλληλα και ανεξάρτητα από τη διαδικασία την οποία ακολουθεί η Γαλλική Αρχή για τις αερομεταφορές. Ήδη έχουν αναλυφθεί κάποιες δράσεις. Η ΕΑΣΑ στις 27 Μαρτίου εξέδωσε ε, ένα νότις ασφαλείας για τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν στην περίπτωση κατά την οποία εγκαταλείπει το κόκπιτ ο κυβερνήτης ή ο συγκυβερνήτης πρέπει να υπάρχει ένα άλλο μέλος ε, του πληρώματος μαζί με τον εναπομείναντα. Εφαρμόζεται πλέον και υποστηρίζεται και από το κοινό. Η Task Force θα επανεξετάσει τις συστάσεις αυτές, όπως επίσης και τις συστάσεις για την ιατρική καταλληλότητα, το ψυχολογικό screening στην αρχή της σταδιοδρομίας και την παρακολούθηση της συμπεριφοράς των κυβερνητών κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας, ε, προβλήματα ανταλλαγής ιατρικών πληροφοριών και φακέλων ιατρικής κατάστασης ανάμεσα σε διαφορετικές αρχές. Η Task Force επίσης θα ελέγχει την κατανάλωση ιατρικών ουσιών και αλκοολούχων ποτών νομίζουμε ότι θα ολοκληρωθεί η πρόταση τον μήνα Ιούλιο και οι συστάσεις της θα ακολουθήσουν προς τον Επίτροπο Μπούλτς. Εμείς εμπιστευόμεθα τους κυβερνήτες του αεροσκάφους και απαιτείται ένα σύστημα ασφαλές το οποίο θα τεκμηριώνει την εμπιστοσύνη αυτή. Το σύστημα αυτό ε, θα γίνεται αντικείμενο διαχείρισης και από τις ίδιες τις επιχειρήσεις και θα βοηθά τους πιλότους να αντιμετωπίζουν με υπεύθυνο τρόπο όποια προβλήματα ψυχολογικά μπορεί να παρουσιάσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και προς όφελος κυρίως των επιβατών. Αυτό το οποίο ονομάζουμε ανθρώπινος παράγων είναι σήμερα κάτι το οποίο ε, είναι καθοριστικό για τη βελτίωση των αερομεταφορών. Αν κάτι συμβεί κατά τη διάρκεια της πτήσης, είναι κάτι το οποίο μπορεί να διορθωθεί και να ανακτηθεί μόνο από τους κυβερνήτες και θα πρέπει να είναι πάντα ικανοί να το κάνουν αυτό, θα είναι εκπαιδευμένοι και σε καλή κατάσταση. Επί τη βάση λοιπόν των προκαταρκτικών αποτελεσμάτων και επί τη βάση των συστάσεων, όπως επίσης και επί τη βάση των συστάσεων τις οποίες σύντομα θα λάβουμε από την Task Force της οποίας ηγείται η ΕΑΣΑ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι διατεθειμένη να αναλάβει τις κατάλληλες δράσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την διασφάλιση της ασφάλειας των Ευρωπαίων επιβατών και των Ευρωπαίων αερομεταφορέων. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κι. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα συμπληρώσω ουσιαστικά αυτά τα οποία είπε ο Φιλίπ Κορνέλιους. Θα δώσω κάποιες περισσότερες λεπτομέρειες για το τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Μετά από την τραγωδία της German Wings. Και θα σας δώσω και κάποιες επιπλέον τεχνικές λεπτομέρειες για τις ενέργειες τις οποίες μέχρι σήμερα έχουμε προβεί. Λοιπόν, εδώ είναι κάποια στοιχεία τα οποία ήδη γνωρίζετε κάποια δεδομένα για το ατύχημα δηλαδή. Πτήσεις από τη Βαρκελόνη στο Ντίσελντορφ, 144 επιβάτες, 6 πλήρωμα. Αριθμός του αεροσκάφους DAIPX Α320-200 συνετρίβει στις Γαλλικές Άλπεις 100 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης της Νίκαιας. Όπως είπε ο Φίλιπ προηγουμένως, ε, της έρευνας ηγείται η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και Ασφάλειας των Αερομεταφορών, η BEA. Ε Εδώ βλέπετε κάποια δεδομένα τα οποία είναι δημόσια πλέον. Να σας θυμίσω λίγο ε, τα στάδια τα οποία οδήγησαν στο ατύχημα με βάση την ανάλυση των καταγραφέων που βρίσκονται στο εσωτερικό του αεροσκάφους. Όλα συνέβησαν σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, συνολικά μικρότερο των 9 λεπτών. Όπως βλέπετε στη συγκεκριμένη διαφάνεια, λίγο πριν από τις 9 και 30, το αεροσκάφος έφτασε στο ύψος πτήσης των 38.000 ποδών και βλέπετε στη συγκεκριμένη διαφάνεια τους αριθμούς με κόκκινο το κόκκινο χρώμα είναι η πραγματική πορεία του αεροσκάφους. Βλέπετε ότι το σημείο 3 είναι το σημείο κατά το οποίο ο κυβερνήτης εγκαταλείπει το κόκπιτ και μέσα σε 10 δευτερόλεπτα αυτό ακολουθείται από μια συγκεκριμένη ενέργεια του συγκυβερνήτη να επιλέξει ύψος πτήσης στο ελάχιστο δυνατό δηλαδή στο επίπεδο της επιφανείας του εδάφους. Βλέπετε αυτό, την μπλε γραμμή. Εκεί επελέγει, κάτω από το σημείο 4 δηλαδή, το χαμηλότερο δυνατό επίπεδο πτήσης. Αυτό το οποίο αξίζει επίσης να δει κανείς, είναι ότι στα σημεία 5 είναι η στιγμή κατά την οποία η ταχύτητα του αεροσκάφους έχει πλέον αυξηθεί από 273 κόμβους σε 308 κόμβους. Στη συνέχεια βλέπετε την αλληλουχία διαφόρων συμβάντων, παρεμβαίνει σαν παράδειγμα ο έλεγχος ενέργειας κυκλοφορίας, ζητά από το κόκπιτ να δηλώσει τις προθέσεις του. Δεν δίδεται απάντηση. Στο σημείο 7 ακούγεται ένα κουδούνι αυτό σημαίνει ότι ζητείτε είσοδο στο κόκπιτ. Μετά από το αίτημα αυτό η ταχύτητα έχει αυξηθεί ακόμα περισσότερο και έχει φτάσει τους 350 κόμβους. Αμέσως μετά ακούγονται ήχοι χτυπήματος στην, ε, πόλη, στην πόρτα του ε, κόκπιτ δυνατά χτυπήματα στο σημείο 11 της αλληλουχίας και στο σημείο 12 φυσικά ακούγεται το σύστημα να προειδοποιεί για την εγκύτητα του εδάφους. Ζητά το σύστημα ε, να ανυψωθεί το ράντερ του αεροσκάφους ε, έτσι ώστε να ανακτήσει ύψος. Φυσικά αυτό είναι απλά η περιγραφή της αλληλουχίας των συμβάνων που οδήγησαν στην τραγωδία. Την 24η Μαρτίου επιβεβαιώνεται το ατύχημα και ξεκίνησε η διαδικασία έρευνας από πλευρά της Γαλλικής Αρχής. Προβλέπεται στην κοινοτική νομοθεσία να οριστεί η ΕΑΣΑ σαν τεχνικό σύμβουλος της αρμόδιας υπηρεσίας έρευνας. Και την ίδια μέρα, ήδη από το απόγευμα της 24ης Μαρτίου, μπορεί να το ενθυμίστε, ε, βρέθηκε ο πρώτος καταγραφέας φωνής. Στις 25 Μαρτίου οι εμπειρογνώμονές μας πήγαν στην ομάδα που ερευνούσε επιτόπου στο ατύχημα, πήραν μέρος λοιπόν στην έρευνα και προσπάθησαν να βοηθήσουν τους ε, ερευνητές με όποιες πληροφορίες είχαμε. Την 26η Μαρτίου ο εισαγγελέας της πόλης της Μασαλίας ανακοινώνει επίσημα ότι πτώση ήταν σκόπιμη και ότι ο συγκυβερνήτης ήταν αυτός ο οποίος ουσιαστικά κατέριψε το αεροσκάφος. Την επόμενη μέρα, μετά από εντατικές διαβουλεύσεις με τις εθνικές αρχές και με ε, αερομεταφορείς, η ΆΣΑ δημοσίευσε συστάσεις εφαρμογής για τις, για τις ε, εταιρείες μεταφορών να υπάρχουν πάντα δύο άτομα στο κόκπιτ καθ' όλη τη διάρκεια της πτήσης έτσι ώστε να εφαρμοστεί η λεγόμενη αρχή των τεσσάρων οφθαλμών. Δημοσιεύθηκε στην την 27η ε, ε, Μαρτίου. Τώρα πώς εμείς εμπλεκόμεθα στην έρευνα. Προβλέπεται από την κοινοτική νομοθεσία αυτό. Είμαστε όπως είπα σύμβουλος α, ε, της υπηρεσίας της Γαλλικής η οποία ασχολείται με την ανάλυση και την έρευνα εμείς δίδουμε στην υπηρεσία αυτή, στην υπηρεσία BEA, πληροφορίες για το τι έχει γίνει μέχρι τώρα για εκτιμήσεις και αξιολογήσεις κινδύνου για ενισχυμένες ασφάλειας θύρες του κόκπιτ, όπως επίσης και για τους κανονισμούς για την ανικανότητα την οποία μπορεί να παρουσιάσει το προσωπικό πτήσης και τον ιατρικό έλεγχο του συγκεκριμένου προσωπικού. Επίσης δώσαμε ε, και την έκθεση των επιπέδων που πρέπει να τηρούνται σε όλους τους τομείς από πλευράς των γερμανικών αρχών και επίσης ε, δώσαμε και ε, κάποια πρώτα στοιχεία της αρχικής μας προκαταρκτικής έρευνας που δημοσιεύθηκε την 6η Μαΐου. Συνεχίζουμε τη συνεργασία μας με τη Γαλλική Υπηρεσία BEA, ιδιαίτερα στον τομέα των ιατροδικαστικών. Όπως είπε ο Φίλιπ Κορνέλης, δημιουργήσαμε μετά από αίτημα της κυρίας Μπούλτς, της Επιτρόπου Μπούλτς, μια task force η οποία έχει σαν στόχο να εξετάσει τα ευρήματα των γαλλικών αρχών της προκαταρκτικής του έρευνας και η διαδικασία που ακολουθείται είναι ότι εμείς με ένα μικρό αριθμό εμπειρογνωμόνων που συμμετέχουν σε αυτήν την Task Force. Προσκαλούμε άλλους εμπειρογνώμονες οι οποίοι καλούνται να μας βοηθήσουν και μας παρουσιάζουν τις απόψεις τους για διάφορα θέματα, κάθε φορά συγκεκριμένα. Αυτό γίνεται παράλληλα με την ανεξάρτητη έρευνα της ΜΕΑ e στη Γαλλία. Έχουμε μια διαφορετική, ένα διαφορετικό χρονισμό οι έρευνες του Μπέρα απαιτούν ένα με δύο χρόνια για να ολοκληρωθούν. Εξετάζουν πάρα πολύ αναλυτικά όλες τις συστάσεις και όλα τα ευρήματα τα οποία υπάρχουν και τα οποία προβλέπονται για τη σχεδίαση του αεροσκάφου σαν παράδειγμα, τις αλλαγές των κανονισμών, των τεχνικών προδιαγραφών κτλ. Αλλά όπως είπε ο Φιλίπ, εμείς θέλαμε να δώσουμε συστάσεις υψηλού επίπεδου προς την Επίτροπο ε, μέσα πριν από το τέλος του καλοκαιριού. Θα ολοκληρώσουμε την έκθεση αυτή τον μήνα Ιούλιο, ελπίζουμε. Έχετε εδώ τα μέλη της Task Force. Βλέπετε ότι υπάρχουν εκπρόσωποι εμπειρογνωμόνων από εθνικές αρχές πολιτικής αεροπορίας, από επιχειρήσεις, αερομεταφορής, εκπροσώπους της Ένωσης του Συνδικάτου δηλαδή των κυβερνητών, των πιλότων. Έχουμε επίσης εκπροσώπους των αεροϊατρικών κέντρων, δηλαδή ιατρικών κέντρων που ασχολούνται με θέματα αερομεταφορών όπως επίσης και εκπροσώπους επιχειρήσεων και επιχειρήσεων αερομεταφορέων εννοώ τις ιδιατρικές τους υπηρεσίες σαν παράδειγμα. Έχουμε κάποιους επίσης εκπροσώπους των οργανισμών εκπαίδευσης των πιλότων. Έχει σημασία να ελέγξει κανείς τα πρώτα βήματα, τα αρχικά βήματα ε, που ακολουθεί ένας υποψήφιος πιλότος. Πέραν τούτων ε, ε, προσκαλούμε εμπειρογνώμονες που συμμετέχουν σε ορισμένες από τις συζητήσεις τις οποίες κάνουμε. Είχαμε εκπροσώπους από τη δική μου υπηρεσία, την ΕΑΣΑ φυσικά. Έχουμε επίσης εκπροσώπους από το FAA, από την Ομοσπονδιακή Αμερικανική Υπηρεσία. Έχουμε επίσης εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Αεροδιαστημικής Υγείας, εκπροσώπους των Γερμανικών Αρχών γιατί όπως γνωρίζετε και η Γερμανία ξεκίνησε την δική της Task Force για να εξετάσει παρόμοια θέματα και αποφασίσαμε ότι θα ήταν καλό να υπάρξει μια στενή συνεργασία και συντονισμός ανάμεσα στις δύο ομάδες. Έτσι λοιπόν, τι κοιτάει η Task Force αυτή. Αυτό αναφέρθηκε ήδη από τον Φιλίπ. Εξετάζουμε πρώτον τα θέματα των θυρών ασφαλείας του κόκπιτ. Όπως γνωρίζετε, κυρίως εξετάζουμε... Ξέρετε ότι οι θύρες αυτές ε, τέθηκαν σε λειτουργία ε, μετά από την 11η Σεπτεμβρίου. Ε, θέσαμε σε εξέταση τα θέματα ασφαλείας για τις κλειδαριές τους, επίσης άλλα θέματα μέσων και διαδικασιών που χρησιμοποιούνται για να κλειδώσουν οι πόρτες αυτές από το εσωτερικό οι κλειδαριές που απαιτούν ανθρώπινη, ανθρώπινο χειρισμό. Κάναμε επίσης ανάλυση των λεγόμενων ιατρικών ελέγχων, δηλαδή αξιολόγηση ψυχολογικών τεστ, αξιολόγηση αρχική και σε συνέχεια συνεχής των πιλότων, έλεγχος για κατανάλωση αλκοολούχων και ναρκωτικών, το πλαίσιο γενικά που καθορίζει την ιδιότητα του εξεταστή στον τομέα αυτό και πώς μπορούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο να ανταλλάξουμε καλύτερα τα ιατρικά αυτά δεδομένα. Το πιο δύσκολο κομμάτι της εργασίας μας ήταν να προσπαθήσουμε να εξετάσουμε το περιβάλλον εργασίας των πιλότων και το θέμα της κοινωνικής ευθύνης ή της ευθύνης την οποία όλοι θα πρέπει να έχουμε όταν εξετάζουμε τον τρόπο με τον οποίο βλέπει την εικόνα του και το περιβάλλον εργασίας του ο πιλότος. Ιδιότερα όταν έχουν προβλήματα οι πιλότοι υγείας, κατάθλιψης κτλ. Προσπαθούμε δηλαδή να δούμε τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται το σύστημα σήμερα. Πού βρισκόμαστε τώρα σήμερα. Τώρα. Έχουμε λάβει αρκετά στοιχεία από την Ομοσπονδιακή Αμερικανική Υπηρεσία για την καλή κατάσταση των πιλότων, αυτά τα οποία απαιτούνται για να κρυθεί κάποιος κατάλληλος στη ΣΥΠΑ. Ανταλλάσσουμε επίσης πληροφορίες με το BDL, την γερμανική υπηρεσία αεροπορίας. Είναι πολύ ενδιαφέρον να ανταλλάσσουμε στοιχεία με αυτή την υπηρεσία στοιχεία στα οποία, τα οποία χρησιμοποιούμε για να καταλήξουμε προφανώς τα ίδια συμπεράσματα. Η τελική συνάντηση της Tax Force προβλέπεται να γίνει στις 16 Ιουλίου. Έχουμε δύο εβδομάδες ακόμα δηλαδή για, το τελικό, για την τελική σύνταξη και να, να τη στείλουμε μετά, αμέσως μετά στο τέλος του μήνα στην Επίτροπο. Αυτά. Ελπίζω να σας έδωσα κάποια επιπλέον στοιχεία. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ο πρόεδρος Κράμερ, σας ευχαριστώ για τις δύο τοποθετήσεις σας. Εκείνο το φοβερό αεροπορικό δυστύχημα μας ε, συντάραξε και μάλιστα αμέσως μετά στην πρώτη μας συνεδρίαση μετά από το δυστύχημα εκείνο τηρήσαμε ενό λεπτού σιγή για να εκφράσουμε τα συναισθήματά μας απέναντι στη μνήμη των θυμάτων και στις οικογένειες των θυμάτων. Υποστηρίξαμε από την αρχή την Task Force. Είπαμε τα πράγματα αυτά. Το σημαντικό αυτό πρέπει να εξεταστεί σε βάθος. Δεν θέλουμε να επαναληφθούν τέτοια πράγματα και γι' αυτό είμαστε και ιδιαίτερα ευγνώμων γιατί η σύνθεσή σας είναι ευρύτατη. Συμμετέχουν εμπειρογνώμονες από τα πλέον διαφορετικά επίπεδα για να ξεκαθαρίσουμε με ποιον τρόπο συνέβη τελικά το συμβάν αυτό και πώς μπορούμε να αποφύγουμε παρόμοια πράγματα στο μέλλον. Σας ευχαριστώ λοιπόν για τις παρεμβάσεις σας και θα δώσω πρώτα τον λόγο στους συντονιστές, στον συντονιστή Βαντε Κάμπ. Α, όχι, δείχνει κάπου αλλού. Α, Μαριάν Μαρινέσκου. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ για τις παρουσιάσεις σας. Φέρθετε λοιπόν με μια τελική έκθεση. Το ερώτημα είναι πώς θα φροντίσετε να εφαρμοστούν οι συστάσεις σας, να γίνουν υποχρεωτικές δηλαδή, γιατί θα πρόκειται για συστάσεις. Οι αεροπορικές εταιρείες θα ακολουθήσουν τις συστάσεις σας αυτές. Πώς πιστεύετε λοιπόν ότι θα μπορέσετε να θέσετε σε εφαρμογή αυτές τις συστάσεις. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Εκ μέρους των Σοσιαλιστών, Αρτούκ. Ευχαριστώ. Στο όνομα της πολιτικής μου ομάδας, σας ευχαριστώ για τις παρεμβάσεις σας. Είναι δύσκολο να μιλήσει κανείς για το θέμα αυτό. Εξηγήσατε άλλωστε και πώς εκτιλήθηκε το δράμα με αρκετά γλαφυρό τρόπο. Κατά την κρίση μου, όπως είπε και ο Πρόεδρος, δεν πρέπει να βιαστούμε. Πρέπει πραγματικά να φροντίσουμε από τα πορίσματα που συλλέγεται εσείς και άλλοι να καταλήξουμε στα πιο στέρεα συμπεράσματα. Βεβαίως λέμε πάντα ότι 100% ασφάλεια δεν μπορεί να υπάρξει. Όμως μπορούμε να κάνουμε προσπάθεια και για ορισμένους τομείς μιλήσατε η πόρτα του πιλωτηρίου. Τι θα γίνει με την ασφάλεια της πόρτας του πιλωτηρίου. Τι θα κάνουμε με τις ιατρικές εξετάσεις. Και αλκοόλ και ναρκωτικά αλλά και ψυχολογικά τεστ. Αυτά που είπατε μου φαίνονται λογικά. Δεν νομίζω όμως ότι μπορούν να αποτελέσουν πανάκια. Γνωρίζουμε ότι στην αρχή της εκπαιδεύσεως γίνεται μια σε βάθος ιατρική εξέταση του προσώπου. Με ενδιαφέρει για να θέσω ερώτηση ταυτόχρονα και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εάν είναι δυνατόν να συζητηθεί να γίνει μια τυποποιημένη διαδικασία εξετάσεων η οποία να γίνεται και να επαναλαμβάνεται τα τακτά διαστήματα. Τονίζω και πάλι ότι δεν μπορεί να αποτελεί πανάκια και η ΕΑΣΑ και η Κομισιόν είπατε και εάν τα αποτελέσματα των ερευνών μου είναι σωστά υπάρχουν ήδη υποστηρικτικά προγράμματα για πιλότους που συνεργάζονται στενά σε peer interaction programs αυτά τα πρόσωπα δηλαδή συνεργάζονται με τις αρχές το ερώτημα είναι αν και από την εργοδοτική πλευρά μήπως θα πρέπει να γίνει υποχρεωτικό για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με την έννοια να νομοθετηθεί. Εξάλλου μου φάνηκε, μου σωστό ότι πολλές αεροπορικές εταιρείες ήδη από την επόμενη μέρα θέσπισαν την αρχή των τεσσάρων ματιών, δηλαδή του δεύτερου προσώπου μέσα στο, στο Έμαθα όμως ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε το εφαρμόζουν ήδη αυτό από καιρό. Θέλω να μάθω λοιπόν αν τώρα αυτή η διαδικασία ισχύει, είναι δεσμευτική και θα είναι δεσμευτική για όλους, δεσμευτική νομοθετικά. Ευχαριστώ, Ρόμπερτ Τζίλε. Ευχαριστώ πολύ τους ειδικού για τις παρουσιάσεις σας, τα σχόλιά σας. Για μας που είμαστε πολιτικοί είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε τι συστάσεις θα έχουμε. Εσείς ως εμπειρογνώμονες καταλαβαίνετε ότι οι θύρες ασφαλείας ήταν ένα μέτρο ασφάλειας μετά την 10η Σεπτεμβρίου. Και τελικά μας οδήγησε σε μια διαφορετική κατάσταση, αυτή που συζητάμε σήμερα. Πώς λοιπόν μπορείτε να διασφαλίσετε ότι οι συστάσεις σας, πολιτικοί είμαστε και το ρωτάμε αυτό, δεν θα, οδηγήσει, δεν θα οδηγήσουν σε μια άλλη επικίνδυνη κατάσταση. Κατά τα άλλα, στηρίζουμε απόλυτα το έργο σας. Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Κύριε Βλυπάου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ πολύ τους δύο προσκεκλημένους μας για τις εξηγήσει τους. Αυτό που είναι σαφές είναι ότι οι τρομοκράτες, οι ομάδες τρομοκρατών τελικά μας προλαμβάνουν. Είμαστε κανονικοί πολίτες ή πολιτικοί και έχουμε την αίσθηση ότι πάντα φτάνουμε αργά. Και αυτό συμβαίνει γιατί βέβαια είναι πάρα πολύ δύσκολο σήμερα να διασφαλίσουμε 100% προστασία. Χαίρομαι πάντως που σε αυτή την ομάδα εργασίας εξετάζεται και το θέμα της κατάρτισης εκπαίδευσης και τα ιατρικά ζητήματα, πώς συνοδεύουμε τον πιλότο, την ασφάλεια στο πιλωτήριο, αλλά και μέτρα που μπορούν να ληφθούν στο μέλλον. Δεν αναφερθήκατε και δεν ξέρω αν είναι δικό σας θέμα, αλλά θέλω να σας ρωτήσω το εξή. Αυτό το ατύχημα οδήγησε σε πολλά θύματα που χρειάζονται βοήθεια, είτε οικογένειες των αποθανόντων, είτε οι τραυματίες. Τους επόμενους μήνες, για να μην πω και χρόνια μετά, χρειάζονται βοήθεια ψυχολογική, τα θύματα και πολλές φορές και στις δικητικές τους διαδικασίες, γιατί είναι υποχρεωμένοι να περάσουν από αυτές. Υπάρχει κάτι σχετικό στην Ευρώπη. Είπα, δεν ξέρω αν είναι δικό σας θέμα, αλλά νομίζω ότι δεν είναι δυνατόν η Επιτροπή μας να μην το αναφέρει και να μην αναφερθούμε και στα δικαιώματα των θυμάτων και των οικογενειών τους. Έχετε συζητήσει καθόλου αυτό το θέμα. Γνωρίζετε μήπως ποια είναι η κατάσταση των οικογενειών των θυμάτων. Είχαν κάποια βοήθεια. Ζήτησαν κάποια βοήθεια. Και τέλος, να μπορούμε να πούμε ότι οι οικογένειες αυτές βοηθούνται. Γνωρίζουμε τις ανάγκες τους και φροντίζουμε να τις καλύψουμε. Σας ρωτάω λοιπόν μήπως θα έπρεπε να συμπεριλάβετε σε αυτήν την task force και κάτι σχετικό με την εφαρμογή των οδηγιών ή των πρωτοκόλων που υπάρχουν για τη βοήθεια στα θύματα. Ευχαριστώ. Λουίς Τεγκράντες. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Είναι προφανές ότι όλοι έχουν την αίσθηση ότι το θέμα της ασφάλειας των αεροπλάνων της αεροπορίας είναι κάτι απαραίτητο για να έχουμε ασφάλεια ακριβώς αεροπορικές μεταφορές. Και το σοβαρό είναι ότι αυτό το τελευταίο τύχημα που συζητάμε οφείλεται σε ένα μέτρο το οποίο είχαμε λάβει πριν από μια προηγούμενη τρομοκρατική ενέργεια. Δηλαδή δεν πρόκειται για κανένα εξωτερικό παράγοντα, πρόκειται για έναν εσωτερικό παράγοντα. Αυτό λοιπόν που ζητάω είναι η ενέργεια ασφάλεια να αντιμετωπίσετε συνολικά. Στους καιρούς που ζούμε η ασφάλεια έχει την ίδια αξία με την ελευθερία. Καθημερινά κάτι γίνεται από εξτρεμιστές, ριζοσπαστικούς, τόσα και τόσα πράγματα. Δεν υπάρχει μηδενικός κίνδυνος. Εδώ έχουμε εκπονήσει διάφορες εκθέσεις πρωτοβουλίες και εγώ ήμουνα εισηγητής και άλλοι για μέτρα. Καταλήγουμε σε σαφή συμπεράσματα όσον αφορά τα αεροδρόμια και τα λοιπά. Και τα αεροδρόμια παίρνουν χρήματα για να κάνουν νέα μέτρα, να εφαρμόζουν νέα μέτρα στην ενέργεια ασφάλεια, κάτι αναγκαίο. Αυτή η task force τώρα θα ήθελα να αφιερώσει λίγο χρόνο, όχι μόνο σε αυτό το συγκεκριμένο ατύχημα, αλλά να λάβει υπόψη τη συνολική αντιμετώπιση της ασφάλειας. Δεν το λέω έτσι ελαφρά. Είναι πράγματα που συμβαίνουν συνέχεια. Υπάρχει τεχνολογία που μπορεί να εφαρμοστεί. Είναι θέμα κόστους το ότι θα εφαρμόσουμε. Ήρθε η ώρα λοιπόν το κόστος αυτό να το αναλάβουμε. Και είναι αναγκαίο οι χώρες μέλη να εμπλακούν, να αναλάβουν το βάρος που πέφτει σε αυτές. Ποτέ δεν θα μπορούμε να προβλέψουμε βέβαια τα πάντα, αλλά μπορούμε να προσφέρουμε περισσότερα στην ενέργεια ασφάλεια για να προβλέψουμε όσα μπορούν να προβλεφθούν, πολύ περισσότερα δηλαδή από όσα σήμερα. Ελπίζω η Task Force δηλαδή να ασχοληθεί και με αυτό και στα συμπεράσματα να συμπεριλάβει κάτι και για το θέμα που ανέφερα. Και έπειτα δεν φτάνουν οι συστάσεις. Χρειάζεται συγκεκριμένη νομοθεσία. Ε, τις μελέτες που έχουν γίνει, από την εμπειρία που έχουμε, να καταλήξουμε σε νομοθετικά μέτρα, να περάσουμε από τις συστάσεις στην επιβολή δημοκρατικά νόμιμα ε, διατάξεων τέτοιων που να ε, καταλήγουν στους στόχους που θέλουμε να πετύχουμε. Ευχαριστώ. έχω γράψει και το δικό μου όνομα. Όντως η αρχή των δύο προσώπων στο πιλωτήριο ισχύει όντω στις ΗΠΑ Πολιτείες αλλά εκεί έχουν και διαφορετικές συνθήκες ασφαλείας. Με ενδιαφέρει τώρα αυτή η αρχή ως εξή. Δύο πιλότοι μέσα στο πιλωτήριο και εφόσον είναι κλειδωμένη η πόρτα δεν γίνεται να επαναληφθεί κάτι τέτοιο παρά μόνο εφόσον συμφωνούν και οι δύο. Το άλλο, το άλλο είναι το τι γίνεται με το ιατρικό απόρριτο. Βεβαίω είναι σημαντικό το ιατρικό απόρριτο, αλλά πρέπει να υπάρχουν και εξαιρέσει για τους γιατρούς όταν διατάσσουν κάποιον να απόσχει από την διεύθυνση του αεροσκάφους. Μπορείτε να απαντήσετε ερωτήσεις αυτές. Μάλιστα. Ευχαριστώ όλους και όλους για τις πολύ συγκεκριμένες ερωτήσεις. Μαρινέσκου πρώτα. Συστάσεις και εφαρμογή τους. Μα εξαρτάται από τις συστάσεις τις οποίες θα καταλήξουμε. Ορισμένες μπορεί τελικά να οδηγήσουν σε αλλαγές των δεσμευτικών κανόνων. Αυτό δεν είναι αναγκαστικό όμως. Μπορεί να υπάρξουν και συστάσεις που προωθούνται και τις οποίες ακολουθεί η βιομηχανία ή ο κλάδος τέλος πάντων ε, εθελοντικά όπως η αρχή των τεσσάρων ματιών που ακολουθείται τώρα εθελοντικά από όλο τον κλάδο. Ερτούγκ. Τακτικές ε, ιατρικές εξετάσεις, peer support program. Αυτά τα έχουμε συζητήσει στην Task Force, δεν έχουμε καταλήξει όμως ακόμα σε τέτοια συμπεράσματα. Δύο άνθρωποι στο πιλοτήριο και η πρακτική που ακολουθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι υποχρεωτική η πρακτική αυτή. Την ακολουθούν πολλές αερογραμμές ως μία λύση. Δεν συνδέεται όμως με μια προσπάθεια πρόληψης τέτοιων συμβάντων, αλλά έχει σχέση με τον χειρισμό της πόρτας. Οι περισσότερες ευρωπαϊκές αερογραμμές έχουν προτιμήσει μια τεχνολογική λύση, δηλαδή ένα κλειστό κύκλωμα τηλεοράσεως όπου βλέπει κανείς από το πιλωτήριο ποιος ε, βρίσκεται μπροστά στην πόρτα. Επομένως είναι θέμα το οποίο έχει σχέση με την ασφάλεια. Ο κύριος Ζήλε, η ισορροπία μεταξύ safety και security των δύο μορφών της ασφαλείας. Θα μιλούμε δηλαδή για την πόρτα του πιλωτηρίου. Βεβαίως γνωρίζουμε ότι υπάρχει συνένεση στον κλάδο αλλά και στους ρυθμιστές ότι η πόρτα του πιλωτηρίου εξακολουθεί, μια ενισχυμένη δηλαδή η πόρτα πιλωτηρίου εξακολουθεί να αποτελεί μια ουσιώδη απέτηση και όντως έχει εξυπηρετήσει το σκοπό της τα τελευταία δέκα χρόνια. Ε, υπάρχει λοιπόν μεγάλη ε, βεβαιότητα σχετικά με αυτό. Η κυρία Ουμπάου ε, μίλησε για τις οικογένειες. Βέβαια, είναι σπάνιο φαινόμενο πλέον στην Ευρώπη να έχει κανείς τέτοια μεγάλα τραγικά ατυχήματα και βέβαια πρέπει να γίνεται κάθε προσπάθεια για να αντιμετωπίσει τις ανάγκες των επιβιώ, επιζώντων. Αυτά βέβαια τα αναλαμβάνουν κυρίως οι χώρες μέλη. Έχουμε πάντως και σε ευρωπαϊκό επίπεδο συνεργασία μέσα σε ένα δίκτυο που λέγεται ΕΝΚΑΖΙΑ και είναι συνεργασία των ερευνητών ασφάλειας και εκεί υπάρχει και μια πτυχή ενίσχυσης των επιζώντων. Είναι βέβαια σπάνια τα συμβάντα αυτά. Αυτό που κάνουμε όμως είναι να ενισχύουμε τις διάφορες χώρες μέλη να διδάσκονται η μια από τα παθήματα της άλλης. Υπάρχουν και κάποιες απαιτήσει, για παράδειγμα οι οικογένειες θυμάτων έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν πληροφορίες στη διάρκεια της ερεύνης. Οι ερευνητές δηλαδή προσπαθούν να ενημερώνουν τις οικογένειες πριν δημοσιεύσουν τις εκθέσεις τους. De Grandes Pasqual, ε, υπενθύμησε άλλο επεισόδιο το οποίο θυμούμαι εγώ καλά και ζητεί μια ολιστική προσέγγιση και εξισορρόπηση θεμάτων ασφάλειας από ατυχήματα και ασφάλειας από τρομοκρατικές ενέργειες. Βεβαίως χρειάζονται περαιτέρω βελτιώσεις της ασφάλειας. Βρισκόμαστε τόσο σε μια διαδικασία επανεξέτασης των βασικών κανονισμών ασφάλειας 216 του 2008 για να τον προσαρμόσουμε στις σημερινές προκλήσεις και ελπίζουμε να μπορέσουμε να κάνουμε πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, μέχρι τέλους του έτους. Ο κ. Κράμερ τέλος μίλησε επίσης για την αρχή των δύο προσώπων μέσα στο πιλωτήριο, για το ιατρικό απόρριτο, βεβαίως είναι ένα θέμα το οποίο μας έχει απασχολήσει πολύ. Η πρόσβαση δηλαδή σε ιατρικές πληροφορίες. Την τάσκο την απασχολεί πολύ αυτό. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος ε, εσείς κύριε τώρα. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ που εκφράσατε το σεβασμό σας για τις ε, εργασίες της Task και δεν παρενέβητε στα θέματα τα τεχνικά. Συμπληρώνοντας αυτά τα οποία εξήγησε ο Φιλίπ, να πω ότι όλα αυτά, αυτό το οποίο δείχνουν και το είπατε κιόλας, ότι η ασφάλεια δεν ε, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με διαφορετικό τρόπο από τα συγκεκριμένα μέτρα τα οποία θα πρέπει να λαμβάνονται κάθε φορά. Πιστεύουμε ότι οι απαιτήσει σε επίπεδο λήψης μέτρων για τις πόρτες των κόκπιτ είναι κάτι το οποίο μπορεί να δημιούργησε κάποιους κινδύνους ασφαλείας γενικότερα. Και αντίστροφα, η επιρροή δηλαδή αρνητική του safety στο security και του Μπαλίν. Είναι λοιπόν σαφές ότι οι ατέλειες που υπάρχουν στη σχεδίαση και στη χρήση των θυρών αυτών ασφαλείας δημιουργούν προβλήματα ασφάλειας. Πρέπει εμείς λοιπόν να δούμε το θέμα σφαιρικά και να αντιμετωπίσουμε και το θέμα των μέτρων ασφαλείας και γενικότερα την ασφάλεια και τους κινδύνους τους οποίους αντιμετωπίζει συνολικά. Ένα από τα θέματα στα οποία αναφερθήκατε είναι ο κανόνας των τεσσάρων οφθαλμών όπως είπα. Εμείς εξετάζουμε το ποιες θα είναι οι συστάσεις. Θα πρέπει να είναι υποχρεωτικές. Γνωρίζουμε ότι στη ΣΥΠΑ κάτι τέτοιο δεν είναι υποχρεωτικό. Συνίσταται απλά, όπως το είπε ο Φιλίπ. Γνωρίζουμε επίσης ότι υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες το κόκπιτ είναι τόσο μικρό που είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπει κάποιος ε, ε, από το υπόλοιπο πλήρωμα και να μην καθίσει στη θέση του συγκυβερνήτη. Αν κάποιος, άνδρας ή γυναίκα, καθίσει στην καρέκλα του συγκυβερνήτη, αυτό μπορεί με τη σειρά του να δημιουργήσει προβλήματα ασφαλείας. Πρέπει λοιπόν να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να λάβουμε υπόψη μας όλα αυτά τα λειτουργικά προβλήματα και τους λειτουργικούς προϋπολογισμούς έτσι ώστε να μεγιστοποιήσουμε τα θέματα ασφαλείας γιατί μερικές φορές το να υπάρχει μια πάρα πολύ δεσμευτική αν θέλετε διακανονιστική ρύθμιση μπορεί να δημιουργεί προβλήματα. Είναι ένα από τα θέματα το οποίο θα πρέπει να εξετάσουμε. Δεν νομίζω ότι θα μπορέσουμε ποτέ να είμαστε σε θέση να επιβάλλουμε στους παθολόγους να δίδουν πληροφορίες για την υγεία του ασθενούς τους είτε σε μία αρχή είτε στον εργοδότη. Δεν υπάρχουν τέτοιοι κανόνες που να υποχρεώνουν ή οδήποτε μέλος του ιατρικού επαγγέλματος να παραβεί τους κανόνες διοντολογίας του. Δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε την πορεία αυτή. Αυτό το οποίο όμως μπορούμε να κάνουμε είναι στα πλαίσια των εξεταστών για την κατάσταση, την σωματική των πιλότων και την ψυχολογική των πιλότων, πώς μπορεί να υπάρξει δυνατότητα ανταλλαγής κρισίμων πληροφοριών, στοιχείων πληροφοριών και ενημέρωσης, όταν θεωρείται ότι υπάρχει κίνδυνος. Ξέρετε ότι στην Ευρώπη μπορεί να μεταφέρουν την άδειά τους οι πτάμενοι από τη μία χώρα στην άλλη. Και γι' αυτό θα πρέπει οι πληροφορίες που συνοδεύουν την άδεια αυτή να είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες, κάτι το οποίο δεν ισχύει σήμερα. Τώρα για τα προγράμματα υποστήριξης στο πτυτικό προσωπικό. Υπάρχουν τέτοια προγράμματα στο εσωτερικό ορισμένων αερομεταφορέων, από ό,τι γνωρίζουμε είναι χρήσιμα, δημιουργούν ένα πλαίσιο, ένα περιβάλλον, μέσα στο οποίο οι πιλότοι μπορούν να υποστηριχθούν και να πάρουν συμβουλές από τους ομολόγους τους έτσι ώστε να μειώσουν το βάρος το οποίο φέρουν. Θα πρέπει να δούμε αν κάτι τέτοιο έχει άμεση σχέση με το είδος της οργάνωσης όπου διεξάγεται ή μπορούμε να γενικεύσουμε αυτούς, αυτές τις ε, μεθόδους. Θα το καταστήσουμε υποχρεωτικό, θα δώσουμε μια λεγόμενη ισχυρή σύσταση. Τι ακριβώς θέλουμε να κάνουμε. Είναι ευαίσθητα τα θέματα αυτά. Πάντως τελικά έχει δίκιο ο κύριος Μαρινέσκου όταν λέγει ότι το ερώτημα είναι με ποιο τρόπο θα μπορέσουμε οι συστάσεις τις οποίες κάνουμε να απαντηθούν, να εφαρμοστούν, συγγνώμη, στην Ευρώπη. Και ένας από τους τρόπους είναι οι σκληρές νομοθετικές ρυθμίσεις, αλλά μερικές φορές μέσω της δημιουργίας νέων δεσμεύσεων δημιουργούμε και προβλήματα. Ίσως θα πρέπει να δημιουργήσουμε ε, κίνητρα για τη βελτίωση του πολιτισμού επιδίωξης ασφάλειας για τις πτήσεις και να βρούμε κίνητρα επίσης για την έβρεση των σωστών μεθόδων εκπαίδευσης και αξιολόγησης. Τώρα για, την τελευταία ομιλήτρια η Task Force δεν θα εξετάσει θέματα αποζημίωσης και κάλυψης του τραύματος των οικογενειών. Εμείς είμαστε μια υπηρεσία ασφαλείας εξετάζουμε τα θέματα ασφαλείας. Έχω πάρει μέρος σε πολλές τελετές για τα θύματα. Βιώνουμε όλη την τραγωδία στην Ιατσά και εκφράζουμε τη θλίψη μας για την κατάσταση στην οποία βρέθηκαν πρώτα απ' όλα τα θύματα βέβαια και οι οικογένειές τους στη συνέχεια. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε τίποτα γύρω από αυτό. Είμαστε αυστηρά υπηρεσία ασφαλείας και ασχολούμεθα μόνο με αυτό. Η Task Force δεν θα ασχοληθεί με τα θέματα αποζημίωσης των οικογενειών των θυμάτων. Είναι ένας τομέας στον οποίο πάντως σίγουρα υπάρχει ανάγκη να συνεχιστούν οι συζητήσεις και να προσπαθήσουμε να βρούμε κοινέ δράσεις. Λοιπόν, αυτά. Νομίζω ότι έδωσα απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις. Ο Πρόεδρος Κράμερ, σας ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση, για την απάντηση των ερωτήσεων. Βεβαίως είναι δυσχερής η κατάσταση. Αναμένουμε την πλήρη έκθεση της Task Force, την οποία θα δημοσιεύσετε, θα μας υποβάλλετε μάλλον τον Ιούλιο ενδεχομένως να μπορέσουμε να τα ξαναπούμε. Ελπίζουμε δε ότι τα συμπεράσματά σας θα οδηγήσουν σε συστάσεις που θα αποτρέψουν ή οδήποτε παρόμοιο ενδεχόμενο στο μέλλον. Σας ευχαριστώ και πάλι. Ja, wir kommen dann zu unserem nächsten Ερχόμαστε στο επόμενο θέμα, δηλαδή την συζήτηση περί κρατικών επιχορηγήσεων στον τομέα των μεταφορών. Ω γνωρίζετε, παίζει σημαντικό ρόλο η, κρατική, η ε, πολιτική επιχορηγήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για παράδειγμα στα λιμάνια, όχι όμως μόνο εκεί. Συζητούμε συχνά τα διάφορα επίπεδα των διαφόρων τρόπων ε, συγκοινωνιών που έχουν διαφορετική μεταχείριση Βεβαίω, η σχετική πολιτική παίζει ένα σημαντικό ρόλο. Καλώ ήρθατε κύριε Γενικέ Διευθυντά τη Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, κύριε Καρλ Σούκουπ και έχετε το λόγο. Χαίρομαι άλλωστε πολύ που είστε κοντά μας. Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε να έρθω και να σας πω δύο λόγια για τις κρατικές επιχορηγήσεις και τις υποδομές μεταφορών. Δέκα λεπτά έχω στη διάθεσή μου, σωστά. Για δέκα διαφάνειες, ένα λεπτό μία δηλαδή. Ωραία, θα προσπαθήσω να το τηρήσω. Προσπαθούμε να είμαστε αποτελεσματικοί στην Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού. Θα δούμε και εδώ αν θα τα καταφέρουμε. Λοιπόν, τα σημεία κίνησης είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να ευθυγραμμίζεται με τις προτεραιότητες της Επιτροπής Juncker για την απασχόληση και τις υποδομές μεταφορών. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα αυτό, άρα δεν εκπλήσει κανέναν ότι ο έλεγχος κρατικών επιχορηγήσεων συμπεριλαμβάνεται. Τι μπορούμε να προσφέρουμε στη χρηματοδότηση υποδομών μεταφορών από πλευράς του ελέγχου κρατικών επιχορηγήσεων. Το πρώτο είναι ότι δεν ζημιώνονται, δεν ζημιώνεται ο ανταγωνισμός στα διάφορα προγράμματα από τις κρατικές επιχορηγήσεις. Δεύτερον, που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και στο οποίο θα επανέλθω και αργότερα, είναι ότι θέλουμε να αποφύγουμε την υπεραντιστάθμιση, δηλαδή η στήριξη που δίνεται στις υποδομές περιορίζεται στο απαραίτητα αναγκαίο, ώστε οι υποδομές να κατασκευαστούν και να δημιουργηθούν περισσότερες ιδιωτικές επενδύσεις. Αυτό που κάνουμε δηλαδή είναι αυτό που λέμε funding gap analysis, δηλαδή να δούμε τι ποσό λείπει προκειμένου να βοηθήσουμε και περιορίζουμε σε αυτό το επίπεδο μόνο τις κατοικές επιχορηγήσεις. Και το τρίτο είναι να διασφαλίσουμε την πρόσβαση στις ε, υποδομές πολλών διαφορετικών φορέων, να μην υπάρχει δηλαδή μονοπόλιο εκεί και κυρίαρχη θέση. Με δύο λόγια. Μην υπάρχει δεσπόζουσα θέση. Με δύο λόγια λοιπόν. Εδώ πρόκειται για την κοινή λογική. Είναι πολύ σημαντικό η χρηματοδότηση για τις υποδομές, να ξέρουμε ότι δεν έρχεται κυρίως από κρατικές επιχορηγήσεις. Και αυτό είναι κάτι το οποίο επιβεβαιώθηκε και από την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Λάτσιπ Χάλε του 2011 όπου διευκρινίζει ότι εάν μία υποδομή χρησιμοποιείται οικονομικά, τότε η οικοδόμησή της ήδη είναι μια οικονομική δραστηριότητα. Αυτό σημαίνει ότι η χρηματοδότησή της έρχεται και ακολουθεί τους κανόνες των κρατικών επιχορηγήσεων. Αυτή είναι η απόφαση λοιπόν, η πρώτη, αλλά υπάρχουν και άλλες. Αυτό σημαίνει από την άλλη μεριά ότι αν η υποδομή δεν τύχει οικονομικής εκμετάλλευσης, όπως για παράδειγμα ένα δημόσιο δικό δίκτυο που χρησιμοποιείται από όλους, τότε χρηματοδότηση αυτής της υποδομής δεν υποβάλλεται στους κανόνες των κρατικών επιχορηγήσεων. Στην πράξη είναι μια ελαστική πολιτική από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχουν πολύ λίγε αρνητικέ αποφάσει στον τομέα αυτό. Και έτσι ε, το ίδιο ισχύει τις αεροπορικές μεταφορές. Και εκεί πρόκειται για τις υπάρχουσες υποδομές όπου εκεί γίνεται επικάλυψη εφόσον υπάρχει και νέα υποδομή κοντά. Αυτό που μας ενδιαφέρει λοιπόν είναι οι κρατικές επιχορηγήσεις να περιορίζονται στο απολύτως αναγκαίο, στο ελάχιστο αναγκαίο. Κυρίως όταν είναι σφιχτός ο προϋπολογισμός και όταν θέλουμε πραγματική προστιθέμενη αξία για τα χρήματα του Ευρωπαίου Φορολογούμενου. Όλα αυτά τώρα προσπαθήσουμε να τα βάλουμε σε ένα σύστημα. Το πρώτο που πρέπει να κοιτάξουμε είναι το εξή. Η υποδομή χρησιμοποιείται για μια οικονομική δραστηριότητα. Ένα αεροδρόμιο, ας πούμε, διόδια, λιμάνι. Εάν όχι, τότε δεν υπάρχει θέμα ε, κρατικών επιχορηγήσεων. Εάν η απάντηση είναι ναι, τότε πρέπει να κοιτάξουμε κατά πόσον οι άλλες προϋποθέσεις, τα άλλα κριτήρια υπάρχουν για να υπάρξει κρατική επιχορήγηση. Τώρα δεν θέλω να σας ζαλίσω με τις ε, λεπτομέρειες, αλλά στο άρθρο 107.1 της Εθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρονται διαφορετικά κριτήρια. Οι κρατικές πηγές, ε, οι επιπτώσεις ε, στον ανταγωνισμό, ας πούμε καθαρά τοπικές υποδομές, η εκμετάλλευση των οποίων δεν επηρεάζει το εμπόριο μεταξύ χωρών μελών, τότε χρηματοδότηση τέτοιων υποδομών δεν περνάει από τους κανόνες κρατικών επιχορηγήσεων. Αν η απάντηση είναι όχι, είμαστε εκτός ελέγχου κρατικών επιχορηγήσεων. Εάν ναι, τότε υπάρχει επιπλέον δυνατότητα να εξετάσει η Επιτροπή. Υπάρχει το τζίμπερ e που σημαίνει ε, ομάδα εξαιρέσεων που ρυθμίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπου μπαίνουν οι προϋποθέσεις. Και αν υπάρχει συμμόρφωση τότε μπορούν να δώσουν επιχορηγήσεις οι χώρες μέλη αλλά πρέπει από πριν έχουν ενημερώσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το άλλο το SGEI πρόκειται για το οικονομικά αποδοτικό. Και εδώ υπάρχει απόφαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν οι προϋποθέσεις και πάλι καλύπτονται, τότε οι κρατικές επιχορηγήσεις δεν πρέπει να κοινοποιηθούν από πριν, εφαρμόζονται από τις χώρες μέλη. Συνεπώς, εάν τα κριτήρια αυτά τηρούνται, τότε μπορεί να δοθεί η κρατική επιχορήγηση χωρίς να περάσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν όμως η απάντηση είναι όχι, τότε πρέπει να γίνει κοινοποίηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς αξιολόγηση. Τι κάνουμε τότε. Τότε κάνουμε μια λογιστική ανάλυση. Κοιτάμε δηλαδή ποιες είναι οι οικονομικές ανάγκες. Ποιο είναι το ποσό που λείπει δηλαδή. Και πρέπει να αποφασίσουμε μέσα σε δύο μήνες μετά την κοινοποίηση. Αυτές είναι οι βασικές αρχές που ισχύουν σε όλους τους τομείς. Εδώ θα περάσω τώρα κάπως πιο γρήγορα σε τέσσερις τομείς υποδομών. Αεροδρόμια, λιμάνια, αυτοκινητόδρομοι και σιδηρόδρομοι. Να σας εξηγήσω ποιοι είναι οι κανόνες που ισχύουν για τα αεροδρόμια. Υπάρχουν κατευθυντήριες γραμμές από το 2014 που έχουν να κάνουν με τις κρατικές επιχορηγήσεις, τις κρατικές επενδύσεις δηλαδή, πάνω από 5 εκατομμύρια, εφόσον είναι επιβάτε στα αεροδρόμια, δεν επιτρέπεται τέτοια επιχορήγηση, γιατί προφανώς τέτοια αεροδρόμια μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις επενδυτικέ τους ανάγκες από μόνα τους. Για αεροδρόμια κάτω από το όριο αυτό, ελέγχουμε διάφορα κριτήρια. Πρόκειται για ένα χρήσιμο σχέδιο, δηλαδή θα στηρίξει την περιφερειακή ανάπτυξη ή θα βοηθήσει να λυθούν προβλήματα εφόσον υπάρχουν. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι δεν πρέπει να υπάρχει επικάλυψη με υπάρχουσες υποδομές, με υπάρχοντα δηλαδή αεροδρόμια. Και υπήρξαν δύο περιπτώσεις όπου η απάντηση από την πλευρά μας ήταν αρνητική. Υπάρχει και το Ghost Airport. Γνωρίζετε και εσείς τις υποδομές αεροδρομίων, τα οποία φτιάχτηκαν με δημόσιο χρήμα και μετά δεν χρησιμοποιήθηκαν ποτέ. Γι' αυτό τα λέμε αεροδρόμια φαντάσματα ή ελάχιστα. Και είναι κάτι το οποίο θέλουμε να αποφεύγουμε στο μέλλον. Είπα επίσης ότι κοιτάμε και το λογιστικό, να δούμε δηλαδή πόσο αναγκαία είναι η χρηματοδότηση κτλ. Όσον αφορά τώρα τη λειτουργική ενίσχυση, αυτή θα συνεχίσει να επιτρέπεται για μικρά αεροδρόμια. Γιατί είναι πιο δύσκολο και τα μικρά αεροδρόμια να καλύψουν το λειτουργικό τους κόστος με ελάχιστα έσοδα. Συνεπώς για πάνω από 3 εκατομμύρια επιβάτες τότε λέμε ότι μπορούν μόνοι τους να τα καλύψουν τα λειτουργικά έξοδα εκείνα που είναι από 700.000 με 3 εκατομμύρια επιβάτε το χρόνο, υπάρχει μια μεταβατική περίοδο για 10 χρόνια προκειμένου να μπορέσουν να προσαρμοστούν στου νέου κανόνε και να αυξήσουν τα έσοδά Και για τα πιο μικρά αεροδρόμια τότε μπορεί να καλυφθεί τουλάχιστον για τα επόμενα 5 χρόνια ε, τα λειτουργικά έξοδα και είπαμε ότι θα ξαναδούμε την κατάσταση το 2018 για να προσδιορίσουμε τους κανόνες για τα επόμενα χρόνια. Ο δεύτερο τομέα στον οποίο θέλω να αναφερθώ είναι οι λιμένε. Εδώ βλέπετε μια χαρακτηριστική δομή, δηλαδή δημόσιες αρχές, οι λιμενικές αρχές, μετά είναι ο πάροχος και στη συνέχεια έχουμε την ε, ναυτιλιακή εταιρεία και τις, ε, και τις δαπάνες που γίνονται. Οι δημόσιες αρχές λοιπόν καταρχήν έχουν ε, το ρόλο να χτίσουν τους ε, πύργους ελέγχου ή τα κτίρια για τα τελωνία κτλ. Μετά υπάρχουν ε, οι λιμενικές εγκαταστάσεις για εμπορικές δραστηριότητες ελέγχουμε όπως και σε άλλες περιπτώσεις κρατικών επιχορηγήσεων, να δούμε αν υπάρχει ο στόχος του κοινού συμφέροντος για να δούμε αν πρέπει να γίνει επένδυση, αν αποτελεί μέρος των διευρωπαϊκών δικτύων, τότε ναι. Και μετά ελέγχουμε και την αναγκαιότητα στους λιμένες, γιατί ίσως να ξέρετε ότι συχνά υπάρχει μεικτή η ένταση, δηλαδή μπορεί να υπάρξει χρηματοδότηση μέχρι ένα ποσοστό. Στα λιμάνια κάνουμε την ανάλυση κόστους πλήρως. Δηλαδή μπορεί να υπάρξει και μέχρι 100% αποδοχή της χρηματοδότησης. Σιδηρόδρομοι τώρα. Η κατάσταση εδώ είναι κάπως διαφορετική. Η γραμμή που ακολουθούμε εδώ είναι ότι η χρηματοδότηση των γενικών υποδομών, δηλαδή της, ε, της σηματοδότησης, που λειτουργεί η ίδια συνδρομική αρχή, που συνήθως είναι δημόσια, δεν θεωρείται κρατική επιχορήγηση, οπότε δεν γίνονται έλεγχοι κρατικής επιχορήγησης. Αν υπάρχει μονοπόλιο για τη λειτουργία των υποδομών αυτών και αν δεν υπάρχει άλλο αντιστάθμισμα. Απ' την άλλη μεριά έχουμε τις εμπορικές υποδομές. Εκεί κάνουμε ένα λογιστικό, μια λογιστική ανάλυση και προσπαθούμε να δούμε κατά πόσο υπάρχουν καλές προκτικές, αν υπάρχει αναγκαιότητα και προσπαθούμε να περιορίσουμε τις επιχορηγήσεις στο ελάχιστο αναγκαίο. Επίσης θέλουμε να υπάρχει και ανοιχτή πρόσβαση σε όλους τους φορείς του δικτύου. Το τελευταίο που θέλω να σας αναφέρω είναι η αυτοκινητόδρομη. Εδώ επιτρέψτε μου να πω ότι η οδεία αυτή είναι εκτός πεδίου κρατικών επιχορηγήσεων. Τι κοιτάμε λοιπόν σε αυτή την περίπτωση, τι ελέγχουμε. Αν υπάρχουν διόδια, επιβάλλονται διόδια διότι η πληρωμή διοδίων θεωρείται μια οικονομική δραστηριότητα. Αυτό που είναι σημαντικό εδώ είναι ότι η κατασκευή και η λειτουργία περνάει από διαγωνισμούς και γίνεται παραχώρηση. Αυτό επιτρέπει να περιορίζεται η επιχορήγηση ή να καταργείται προς τον παραχωρησιούχο. Υπάρχουν διαφορετικές δυνατότητες τώρα για να δούμε κατά πόσο είναι συμβατή μια επιχορήγηση ή όχι. Χρησιμοποιούμε διάφορα κριτήρια. Τη δυνατότητα να οριστεί ένα πρόγραμμα το οποίο να είναι ε, κοινού ευρωπαϊκού συμφέροντος, ας πούμε, να χτιστεί μια γέφυρα, κάτι που έγινε πέρυσι. Και εδώ πάλι προσπαθούμε να περιορίσουμε το ποσό της επιχορήγησης. Συνοψίζοντας λοιπόν στις προηγούμενες διαφάνειες. Οι υποδομές μεταφορών περνούν από έλεγχο κρατικών επιχορηγήσεων εφόσον ε, πρόκειται για μια οικονομική δραστηριότητα. Αν υπάρχει, υπάρχουν διόδια, αν υπάρχει κάποιο τέλος περιορίζουμε την επιχορήγηση αυτή στο των δυνατόν. Ελάχιστες αντικές αποφάσεις έχουν ληφθεί μέχρι τώρα. Γίνονται συζητήσεις με τις χώρες μέλη για τα προγράμματα, τον ορισμό τους, για την οικονομική ανάλυση αν περιορίζεται η επιχορήγηση σε σχέση με το αρχικό μπορούμε να συμφωνήσουμε. Σπάνια έχουμε αρνητικές αποφάσεις. Λαμβάνουμε υπόψη μας τις ιδιαιτερότητες επίσης του τομέα. Δεν έχουμε μια ενιαία αντιμετώπιση για όποια υποδομή και αν πρόκειται. Γνωρίζουμε ότι διαφορετικοί τομείς χρειάζονται διαφοροποιημένη μεταχείριση. Και πρέπει να πούμε Νομίζω ότι τις αποφάσεις τις φέρνουμε, δεν θα έλεγα γρήγορα, αλλά εν πάση περιπτώσει σε λογικό χρονικό διάστημα. Εξαρτάται φυσικά από τις πληροφορίες που έχουμε και από το πρόγραμμα, την ποιότητα του προγράμματος δηλαδή που μας υποβάλλεται. Αυτά ήθελα να σας εξηγήσω. Και από εκεί και πέρα ευχαρίστω να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Ο πρόεδρος Κράμερ, σας ευχαριστώ για την τοποθέτησή σας. Ο κύριος Μάρκους Φέρβερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και πρώτα ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ανάπτυξη του θέματος. Είναι πια σαφές. Βρισκόμαστε άλλωστε στο πλαίσιο της Connecting Europe Facility και εκεί προσφέρουμε και επιδοτήσεις. Είναι σημαντικό λοιπόν να τα γνωρίζουμε αυτά. Επιδοτήσεις που μπορούν να θεωρηθούν ως κρατική επιδότηση. Ε, είναι σαφές λοιπόν ότι οι υποδομές χωρίς την επιχορήγηση του δημοσίου δεν θα τα καταφέρουν. Και τα παρακολουθούμε αυτά βέβαια και στην, στα πλαίσια της εξέλιξης του FSI. Έχω κάποιες αμφιβολίες αν μπορεί το ιδιωτικό κεφάλαιο να αναπληρώσει την ενδεχόμενη έλλειψη ε, της δημόσιας ε, χρηματοδότησης. Εδώ θέλουμε ωστόσο να μάθουμε σήμερα Παίζει σωστά το ρόλο της Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως διαιτητής που καμιά φορά μπορεί να μην είναι δημοφιλής αλλά οφείλει να ε, φροντίζει ώστε να εφαρμόζουν όλοι τους ίδιους κανόνες. Διακόπτεται το, μικρόφωνο του κ. Φέρμπερ. Τώρα τον ακούμε πάλι. Είναι λοιπόν σημαντικό να παίξει το ρόλο αυτό. Δεν έχω βέβαια τίποτε σπουδαίες ερωτήσεις εκτός από το εξής έχουν υποβληθεί κάποιες υποθέσεις και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Υπάρχουν καμιά φορά διαφορέ απόψεων μεταξύ χωρών μελών και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται στον τομέα αυτό και εφαρμόζει και το εργαλείο ρυθμίσεων τις οποίες αυτό αποφασίζει σε ό,τι αφορά τη διαφάνεια. Όπου εκεί το Κοινοβούλιο έχει περιορισμένο δικαίωμα συμμετοχής και οι χώρε μέλη ακόμη έχουν περιορισμένο δικαίωμα συμμετοχή εφόσον μόνο ακούει τη γνώμη τους. Αυτό συμβαδίζει με την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Έχω και μια άλλη ερώτηση. Όχι ευθέω για τις υποδομέ για τη χρηματοδότηση αερογραμμών, που και εκεί υπάρχουν ειδικέ ρυθμίσεις. Εκεί είστε επίσης αρμόδιος εσείς και το τμήμα σας ή πρέπει να ε, ακούσουμε κάποιον άλλο. Ο κ. Σερτούγκ ε, αποποιείται. Καριμαντελή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, Ευχαριστώ και τους εκπροσώπους της Επιτροπής. Θα ήθελα να πω ότι σήμερα υπάρχουν πάρα πολλά περιφερειακά αεροδρόμια τα οποία υπερχρηματοδοτούνται. Και όπως αποδεικνύει η έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου, αδίκως. Πώς μπορείτε να μας διαβεβαιώσετε ότι οι χρηματοδοτήσεις αυτές θα καταστούν αποτελεσματικές. Αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση. Αναφερθήκατε στον έλεγχο. Πώς ελέγχονται οι επιδοτήσεις αυτές και επί τη βάση ποιων κριτηρίων, με ποιο τρόπο θα μας εξασφαλίσετε ότι ε, ε, στην ουσία οι επιδοτήσεις αυτές δεν δίδονται στρεβλά προς ε, ενίσχυση των low cost, των εταιριών χαμηλού κόστους. Όπου υπάρχουν επιδοτήσεις σε περιφερειακά αεροδρόμια, ένα τμήμα πηγαίνει σε αεροπορικές επιχειρήσεις οι οποίες δεν σέβονται τους ισχύοντες κανόνες. Θα λάβετε κυρώσεις σήμερα για εναντίον όλων αυτών των πρακτικών και αυτών ε, οι οποίοι τις φέρουν εις πέρας. Φαντερκάμπ. Πρόεδρε. Οι δύο ερωτήσει μου. Στο θέμα των μεταφορών και στη Λευκή Βίβλο έχουμε το κεφάλαιο εσωτερήκευση του εξωτερικού κόστος. Είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό στον κόσμο μας, η εσωτερήκευση του εξωτερικού κόστους μπορεί να συμπεριλάβει και τις κρατικές επιχορηγήσεις. Έχουμε την πράξη του Μανχάιμου που λέει ότι ε, μπορείς δωρεάν να ανακαινηθείς στο Ρήνο, ποιος όμως κάνει τη συντήρηση του Ρήνου. Τέτοιου είδους οριακές ε, καταστάσεις υπάρχουν. Υπάρχουν ε, λιμένια, λιμάνια που έχουν δωρεάν υποδομές και άλλα που δεν πληρώνουν τέλη. Είναι και αυτό κρατική επιχορήγηση, δεν είναι. Και έρχομαι τώρα στο σιδηροδρόμου. Στο πακέτο το σιδηροδρομικό έχουμε την αναλογία ανάμεσα στην ε, εταιρεία που φροντίζει για το ταξίδι και από την άλλη μεριά έχουμε τη διαχείριση των υποδομών. Στο πακέτο αυτό το σειρονομικό λοιπόν πρέπει να δούμε τι επηρέαζε τι, ποιος επηρέαζε ποιον. Και τρίτον, οι χώρες μέλη ε, πολλές φορές βάζουν τη φαντασία τους ε, να δουλέψει και βρίσκουν άλλους τρόπους κρατικών επιχορηγήσεων. Εσείς φροντίζετε να κυνηγήσετε και αυτές τις περιπτώσεις, δηλαδή κυνηγάτε και αυτές τις δημιουργικές ε, κρατικές επιχορηγήσεις. Ευχαριστώ. Τρεις ερωτήσεις και από εμένα, λέει ο πρόεδρος Κράμερ. Με εξέπληξε λίγο που είπατε ότι λίγα μόνο έργα σε λίγα μόνο έργα ήταν εσφαλμένα τα πράγματα. Πρόσφατα συζητήσαμε τα περιφερειακά αεροδρόμια Κανένα δεν μα είπε ότι είναι εντάξει τα πράγματα από 8 χώρε. Και αυτό με εκπλήσει λίγο που λέτε only a few. Saarbrücken, Zweibrücken. Ε, μικρή απόσταση μεταξύ τους και τα δύο ελληματικά, επειδή όμως είναι σε διαφορετικά ομόσπονδα κρατήδια, Γι' αυτό υπάρχουν δύο αεροδρόμια. Όμως από 23 διεθνή αεροδρόμια στη Γερμανία τα 17 είναι ελληματικά. Αυτά δεν τα περίμενε κανείς. Να τα μάθει. Πρόκειται τώρα για ανεπίτρεπτη η υποστήριξη όταν για παράδειγμα οι αερογραμμές δεν πληρώνουν φόρο επί της κυροζήνης ενώ οι επιβάτες των σιδηροδρόμων πληρώνουν. Έχουμε άλλο κανόνα ότι η μηχανή έλξεως πληρώνει για κάθε χιλιόμετρο που καλύπτει στον σιδηρόδρομο ένα διόδιο. Δεν το πράττουν αυτό τα φορτηγά αυτοκίνητα ή πάντως όχι κάτω από 12 τόνους. Μήπως πρόκειται εδώ για παράνομη επιδότηση που έχει τρομερές επιπτώσεις και ασφαλμένες μάλιστα. Τέλος, για το, ...υπάρχει για τα αεροδρόμια. Είμαι Βερολινέζος. Υπάρχει και ένα αεροδρόμιο το οποίο υποτίθεται ήταν έτοιμο εδώ και τρία χρόνια. Δεν μιλώ τώρα γι' αυτό όμως. Υπάρχουν κάποια αεροδρόμια τα οποία έχουν ιδρυθεί με ιδιωτικά χρήματα. Το αεροδρόμιο του Βερολίνου ωστόσο χρηματοδοτείται από το Ομόσπονδο και από την Ομοσπονδία. Δηλαδή τους χαρίζουν, χαρίζουν στις αεροπορικές εταιρείες την υποδομή. Άλλα αεροδρόμια όμως οφείλουν να τα χρηματοδοτήσουν ήδη. Ή έχουμε και τις low cost airlines που κάνουν κάποια αμφίβολης νομιμότητας, κάποιες αμφίβολης νομιμότητας ε, συμβάσεις με κάποιες περιφέρειες και χρησιμοποιούν διάφορα τρίκ για να εξασφαλίζουν τις επιδοτήσεις. Αυτά τα τρίκ τα αποκαλύπτετε εσείς και τους καλείτε μετά να πληρώσουν, επιβάλλονται κυρώσεις έτσι ώστε να αποτρέπονται στο μέλλον τέτοιες πρακτικές. Εν τέλει θέλουμε βέβαια θεμητό και όχι αθέμητο ανταγωνισμό. Σας ευχαριστώ πολύ και αν θέλετε παρακαλώ απαντήστε τώρα σε ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις. Να αρχίσω με μια γενικότερη δήλωση που καλύπτει νομίζω κάποιες ερωτήσεις. Η πολιτική και το δίκαιο του ανταγωνισμού και κυρίως των κρατικών ελέγχων είναι ένα ε, βαρύ εργαλείο στα χέρια της Κομισιόν. Εμείς είμαστε ο ανεξάρτητος διευθυντής, όπως το είπε σωστά ο κ. Φέρβερ. Είναι λοιπόν σημαντικό όπλο και πρέπει να το χρησιμοποιούμε με προσοχή. Βέβαια δεν μπορεί να λύσει όλα τα προβλήματα το εργαλείο αυτό. Υπάρχει και ο πειρασμός να αντικαταστήσουμε τους υφιστάμενους κανονισμούς με την χρήση των ε, ε, εργαλείων για τον ανταγωνισμό. Βέβαια δεν είναι όλα τέλεια, πρέπει ορισμένα να τροποποιηθούν ή να αλλάξουν. Στις περισσότερες περιπτώσεις η ρύθμιση είναι καλύτερα να υπάρξει παρά επιβολή του δικαίου του ανταγωνισμού. Για παράδειγμα, μιλήσατε για την εξαίρεση από τον φόρο στην κυροζήνη που από όσο γνωρίζω θεσπίζεται με ευρωπαϊκή νομοθεσία. Με συγχωρείτε να σας διακόψω λέει ο πρόεδρος Κράμερ. Όχι, πρόκειται για τη σύμβαση του Σικάγο. Αυτή λέει ότι η κυροζήνη που είναι μέσα στο αεροσκάφος όταν αυτό προσγειώνεται δεν φορολογείται. Κάθε χώρα, άρα και η Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορεί να επιβάλλει φορολογία επομένως. Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως αποφάσισε να μην το πράξει. Και αυτή η απόφαση έχει θεσπιστεί νομοθετικά. Επομένως είναι κάτι το οποίο επιβάλλεται από τον Ευρωπαίο νομοθέτη. Άρα η χώρα μέλος δεν έχει περιθώριο κίνησης ελιγμού. Επομένως η εξαίρεση αυτή δεν μπορεί να βαρύνει την χώρα. Δηλαδή δεν μπορεί η χώρα μέλος να θεωρηθεί υπεύθυνη μη ορθής εφαρμογής της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Υπάρχει και σχετική, υπάρχει και σχετική νομολογία του δικαστηρίου για τους γερμανικούς σιδηροδρόμους το Λουξεμβούργο δηλαδή το δικαστήριο του Λουξεμβούργου είπε ακριβώ αυτό ότι στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει κρατική επιχορήγηση διότι τη σχετική εξαίρεση θεσπίζεται από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Αν θέλετε λοιπόν να λύσετε το πρόβλημα αυτό, νομίζω τότε θα πρέπει να τροποποιήσετε την κείμενη νομοθεσία. Τώρα, να έρθω σε ερωτήσει. Κύριε Φέρβερ. η συμβατότητα προκύπτει από δίκαιο της Κομισιόν. Soft law που είναι δεσμευτικό για την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά υπόκειται στον έλεγχο του δικαστηρίου. Πολλές αποφάσεις μας άλλωστε προσβάλλονται από ανταγωνιστές ή δικαιούχους ενώπιον του δικαστηρίου του Λουξεμβούργου και ορισμένες φορές μας ανακαλούν σε τάξη. Συχνά Επιβιώνεται η ισχύ των αποφασιών μας και είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένο γι' αυτό. Πάντω υφιστάμεθα τον έλεγχο αυτό και κάθε φορά που μας βαλώνει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο το λαμβάνουμε αυτό υπόψη και τροποποιούμε τους κανόνες μας. Σε ό,τι αφορά τις Aviation Guidelines του 2014 και εκεί υπάρχουν κανόνες για την υποστήριξη των αεροπορικών εταιριών από τα αεροδρόμια ώστε οι συμφωνίες μεταξύ airlines και αεροδρομίων ρυθμίζονται σε αυτές τις κατευθυντήρες γραμμές. Και έτσι απαντώ και στην ερώτηση εάν μάλλον πώς μπορούμε να αποφύγουμε να διοχετεύεται βοήθεια στα αεροδρόμια σε low cost carriers. Εφόσον η σύμβαση μεταξύ του αεροδρομίου και της αεροπορικής εταιρείας αποτελεί μια γενικώ θετική προσθέμενη αξία για το αεροδρόμιο, δηλαδή προσφέρει περισσότερα πρόσθετα έσοδα από δαπάνες. Το, δικαστη... το, συγγνώμη, αεροδρόμιο πρέπει να έχει ένα business plan το οποίο να το καθιστά βιώσιμο και τότε μόνο μπορεί να χωρεί εκεί μια συμφωνία με μια αεροπορική εταιρεία. Επιπροσθέτως, για τις βοήθειες αυτές μέσω αεροδρομίων, και εδώ αναφέρομαι και στις κρατικές επιχορηγήσεις προς ε, αεροπορικές εταιρείες οι οποίες βρίσκονται σε δυσχέρειες, μιλούμε εκεί για restructuring, Καμιά φορά λαμβάνουμε θετικέ αποφάσεις, καμιά φορά λαμβάνουμε αρνητικέ αποφάσεις. Εάν η αποκατάσταση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας δεν μπορεί να επιτευχθεί, όπως για παράδειγμα στη Cyprus Air, όπου αναγκαστήκαμε να λάβουμε αρνητική απόφαση διότι σε τέτοια περίπτωση αν δινόταν αυτή η ε, βοήθεια θα επανερχόταν στην ίδια κατάσταση μετά από λίγο καιρό η αεροπορική εταιρεία γιατί δεν μπορούσε να σταθεί από μόνη τα πόδια της. Τώρα, για υπερχρηματοδοτούμενα αεροδρόμια που βρίσκονται σε ανταγωνισμό με άλλα. Γνωρίζω ότι το ελεγκτικό συνέδριο τήρησε πολύ επικριτική στάση απέναντι σε αυτό. Έχει μέχρι τώρα εκδώσει τρει αρνητικέ αποφάσεις, αλλά συνεχίζονται πολλές, εκκρεμούν ακόμα πολλές υποθέσεις. Μετά από τις guidelines του 2014 έχουμε αρχίσει να ξεκαθαρίζουμε τις υποθέσεις μας. Λήφθησαν πολλές αποφάσεις στο δεύτερο εξάμεινο του περασμένου έτους. Μεταξύ αυτών μάλιστα ήταν τρεις, όπως είπα, αρνητικές αποφάσεις. Μία από αυτές αναφερόταν στο αεροδρόμιο Τσφάιμπρουκεν που είπατε προηγουμένως εσείς και το ε, αεροδρόμιο του Ζαρμπρουκεν είναι περίπου 30 χιλιόμετρα μακριά από το Τσφάιμπρουκεν. Παρόμοια κατάσταση βλέπουμε στην Πολωνία, στα αεροδρόμια Κτίνια και Ντάνσκ, και Γκτάνσκ, διότι εκεί δεν βλέπουμε το λόγο να υποστηρίξουμε ένα αεροδρόμιο που βρίσκεται εγγύς άλλου υφιστάμενου ε, αεροδρομίου που έχει χαμηλή ε, χωρητικότητα. Έχει free capacity, έχει δεύτερη χωρητικότητα. Έτσι δεν μετρούν για μας και αυτά τα ε, ομοσπονδιακά επιχειρήματα που προβάλλονται στη Γερμανία όσον αφορά αεροδρόμια τα οποία βρίσκονται σε δύο χωριστά ομοσπονδιακά κρατήδια. Ο υπολογισμός εσωτερικά του κόστους τους. Ποιος είναι υπεύθυνο γι' αυτό. Υπάρχει μια ενδιαφέρουσα συζήτηση η οποία γίνεται και εδώ στα πρέσβη στα πλαίσια της πρότασης κανονισμού για τις υπηρεσίες ε, στους αερολιμένες. Αντίστοιχες σκέψεις λέμε και για το ποιες υπηρεσίες στα αεροδρόμια είναι οικονομικής φύσεως. Αντίστοιχα και στους λιμένες, γιατί όπως είπα πριν, αυτό έχει συνέπειες στην προσπάθεια κατανόησης της φύσης των υπηρεσιών αυτών. Έχουμε στείλει ένα ερωτηματολόγιο σε όλα τα κράτη-μέλη, ρωτώντας τα για τον τρόπο με τον οποίο οργανώνονται στον τομέα αυτόν. Πρέπει να πούμε ότι δεν υπάρχει ομόφωνη αντίληψη των κρατών μέλων για κάποιες από τις υπηρεσίες αυτές και η εμβάθυνση των λιμένων είναι κάτι το οποίο δεν έχει τύχει μίας απάντησης.

των επιχειρήσεων που είναι υπεύθυνα για τους σιδηροδρόμους και για τα δίκτυα. Αυτό το οποίο είναι θετικό είναι το θέμα θετικό, είναι σημαντικό μάλλον, είναι το θέμα της διαφάνειας. Το θέμα της προέλευσης των χρημάτων επίσης, αν υπάρχουν διασταυρούμενες μορφές επιδότησης, Υπάρχουν επίσης και κάποιες, ε, κάποια παραθυράκια τα οποία γνωρίζουμε ότι υπάρχουν και θέλουμε να τα κλείσουμε. Εδώ ε, η έλλειψη διαφάνειας δεν διευκολύνει τους κανόνες αυτούς. Εμείς παρακολουθούμε τα θέματα της δημοσιοποίησης, της δημοσίευσης, ε, παρακολουθούμε τα θέματα των παραπώνων, των αναφορών, επίσης και της γνωστοποίησης των επιδοτήσεων Πολλές φορές οι χώρες δεν είναι ιδιαίτερα συνεργάσιμες ε, στα πλαίσια της ενημέρωσης ε, για την ύπαρξη επιδοτήσεων βοήθειας προς ε, κάποιους τέτοιους οργανισμούς. Συλλέγουμε πληροφορίες και από παραπονούμενους και από ΜΚΟ. Εξετάζουμε προσεκτικά λοιπόν τις ανησυχίες αυτές και την ενημέρωση αυτή. και αν χρειαστεί θα ξεκινήσουμε περισσότερες διαδικασίες για το Βερολίνο τώρα. Δεν είμαι ιδιαίτερα οικείος με την υπόθεση αυτή. Νομίζω ότι εν αρχή χρηματοδοτήθηκε από το κράτος και όχι αυστηρά ιδιωτικά για το συγκεκριμένο αυτό αεροδρόμιο, το Τέγκελ οι περισσότερες αερολιμανικές υποδομές στην Ευρώπη σε κάποια φάση στην ιστορία τους στηρίχθηκαν οικονομικά από το κράτος με δημόσιο χρήμα. Αναθεωρήσαμε κάποιους κανόνες πέρυσι, είπαμε ότι θα υπάρξουν μεταβατικές περίοδοι και σταδιακή εισαγωγή των νέων μέτρων, έτσι ώστε τα αεροδρόμια να μπορέσουν να προσαρμοστούν και να καταστούν βιώσιμα από, ε, από δημόσιες χρηματοδοτήσεις. Κάνουμε διαφορές ανάμεσα στους μεγάλους αερολιμένες που είναι αυστηρά εμπορικές επιχειρήσεις, πρέπει να είναι, και μικρούς αερολιμένες οι οποίοι αντιμετωπίζουν περισσότερες δυσκολίες για την κάλυψη του κόστους, κάτι το οποίο στηρίζει στόχους ανάπτυξης της υπαίθρου περισσότερο ε, και δεν λειτουργεί όπως τα μεγάλα κομβικά αεροδρόμια στην Ευρώπη. Σας ευχαριστώ για την παρέμβαση και βεβαίω για την απάντηση των ερωτήσεων. Πριν έρθουμε τώρα... Α, διακόπτει ο πρόεδρος. Ο κ. Φέρβερ. Συμπληρωματική ερώτηση για τα αεροδρόμια. Έχουμε διάφορα χρηματοδοτικά μοντέλα. Έχουμε χρηματοδοτικά μοντέλα όπου ο, η εταιρεία λειτουργίας του αεροδρομίου λαμβάνει πιστώσεις με εγγυήσει των χωρών μελών. Έχουμε μετά αεροδρόμια που χρηματοδοτούνται ιδιωτικά. Έχουμε αεροδρόμια όπου διαθέτει δωρεάν την υποδομή το κράτος. Μπορώ να σα πω διάφορα μοντέλα Εκεί, εκεί ισχύουν διαφορετικοί όροι ανταγωνισμού, διότι το πρώτο και δεύτερο μοντέλο θα πρέπει να κερδίζει από τα τέλη χρήσεως της υποδομής, ενώ στην τρίτη περίπτωση όχι. Εκεί δεν επιβάλλεται κανένα κόστος στην ε, εταιρεία λειτουργία του αεροδρομίου, έτσι δεν είναι. Κράμερ. Ε, Βεβαίω υπάρχει διαφορά. Για το νέο αεροδρόμιο του Βερολίνου, όχι πλέον το Τέγελ, αλλά για το Σένεφελτ, είχε προβλεφθεί στον αρχικό σχεδιασμό προστασία από το θόρυβο και οι, αυτοί που λειτουργούν το αεροδρόμιο, δηλαδή τα δύο κρατήδια και η Ομοσπονδία, διέγραψαν την ε, προστασία κατά του θορύβου. Τώρα, μετά από προσφυγές των περιοίκων, οφείλουν ε, να προσφέρουν και αυτοί, δηλαδή να, να, να ε, προβλέψουν και αυτή την προστασία κατά του θορύβου. Και τώρα επειδή είναι πιο ακριβό, δηλαδή θα κοστίσει 4 δισεκατομμύρια και όχι 2 δισεκατομμύρια, ζητούν συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι γνώμη έχετε. Έχουν πιθανότητες να λάβουν χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρείτε ότι αυτό είναι δίκαιο. Αυτό έντιμο και δίκαιο, ξέρω εγώ, είναι κάπως ε, λίγο βαλή χαρακτηρισμοί. Μου φαίνεται να είναι γερμανική συζήτηση αυτή, αλλά παρόλα αυτά επιτρέψτε μου να απαντήσω στα αγγλικά. Μιλώ για το αεροδρόμιο του Μονάχου, το οποίο είναι δημόσια χρηματοδότηση. Μαλπένσα στο Μιλάνο επίση, ιδιωτικό αεροδρόμιο. Και το Ζάβεντεμ στο Βέλγιο, απολύτω κρατικό, διατίθεται δωρεάν ω υποδομή. Έχετε λοιπόν και τα τρία παραδείγματα. Ε, με συγχωρείτε, λέει ο Ευρώπη Κομισιόν, δεν είμαι αρνητικά διατεθειμένο κατά τη Γερμανία. Εδώ μιλούμε και για εγγυήσει δανείων. Είναι κρατική επιδότηση. Είναι κρατική επιδότηση. Είτε είναι δημόσιος δανεισμός, είτε είναι ε, ε, εγγύηση. Θεωρούνται και αυτά κρατική επιδότηση. Όπως προσπάθησα να εξηγήσω πριν, από τα μισά του περσινού χρόνου όταν άρχισαν να ισχύουν οι κατευθυντήριες γραμμές, η χρηματοδότηση αεροδρομίων άνω των 5 εκατομμυρίων επιβατών καταρχήν δεν συμβαδίζει με τους κανόνες μας. Ωστόσο τέτοιου είδους επενδύσεις θα πρέπει να, ε, να χρηματοδοτούνται από τα ίδια τα αεροδρόμια. Υπάρχουν βέβαια κάποιες εξαιρετικές περιστάσεις που μας επιτρέπουν να αποκλίνουμε από την πρόβλεψη αυτή, αλλά δεν έχει συμβεί ως τώρα τι ακριβώς επιβάλλουμε τον κανόνα αυτό. Αφενός διότι γνωρίζουμε ότι υπάρχουν διαφορετικά μοντέλα χρηματοδοτήσεως και δεν θέλουμε να προβούμε σε διακρίσεις υπέρ ή κατά των μεν ή των δε. Εάν ένα αεροδρόμιο πληρώνει από μόνο του όλες τις υποδομές ενώ ένα άλλο αεροδρόμιο τις λαμβάνει δωρεάν από το κράτος υπάρχει διαστρέβλωση στον ανταγωνισμού, είναι προφανές. Ιδίω όμως για μικρότερα αεροδρόμια ίσως να είναι αναγκαίο αυτό και μάλιστα ίσως να είναι και προς το δημόσιο συμφέρον να υποστηριχθούν τα αεροδρόμια αυτά. Όμως συμφωνώ μαζί σας ότι τα μεγάλα αεροδρόμια, και νομίζω για αυτά μιλούμε περισσότερο τώρα, δεν θα πρέπει να δίνεται ε, επενδυτική υποστήριξη. Τώρα για το αεροδρόμιο του Βερολίνου και αυτά που είπατε για την επερχόμενη αυτή υπόθεση, δεν θέλω να ε, κάνω εικασίες για μια υπόθεση που μπορεί να τεθεί υπόψη μας στο μέλλον, δεν θέλω να προκαταλάβω την ανάλυση που θα κάνουμε. Έχουμε ωστόσο συζητήσει την υποστήριξη για το αεροδρόμιο του Βερολίνου στο παρελθόν και νομίζω η θετική απόφαση της Κομισιόν για το αεροδρόμιο BER εφόσον αποδειχθεί ότι απαιτούνται πρόσθετα μέτρα είμαι βέβαιος ότι η Γερμανία θα έλθει να μας βρει και να συζητήσει μαζί μας και είμαι βέβαιος θα είναι τότε σε πλήρη συμφωνία με τους όρους του ανταγωνισμού. Βεβαίως θα έρθει η Γερμανία, μα εκεί μιλούμε όμως για 20-25 εκατομμύρια επιβάτες. Είπατε ότι από 5 εκατομμύρια επιβάτες και πάνω δεν υπάρχει πλέον κρατική επιδότηση. Αυτό είναι το ερώτημα. Βέβαια καταλαβαίνω ότι δεν θέλετε να απαντήσετε ακόμα. Αλλά κανονικά αποκλείεται να δοθεί αυτή η επιδότηση. Έτσι είναι. Και τότε όλα αυτά είναι δίκαια και έντιμα. Δεν θα έλεγα ότι δεν μου επιτρέπεται να πω, δεν μπορώ να πω απαντά ο Αρχός Κομισιόν, δεν μπορούμε άλλωστε ω αξιωματούχοι τη Κομισιόν να προκαταλάβουμε τι αποφάσει του Κολεγίου των Επιτρόπων. Σίγουρα πάντω θα είναι μια δύσκολη ε, υπόθεση. Μάλιστα, Σα ευχαριστώ πολύ. Ξεκάθαρα πράγματα και τώρα ξέρουμε όλοι καλύτερα τι συμβαίνει. Σα ευχαριστώ πολύ. Πριν προχωρήσουμε τώρα στο επόμενο θέμα της μεσαίας διατάξεως, το οποίο θα διαξαχθεί και κλεισμένο των θυρών, έχω μια αλλαγή να σα ανακοινώσω εδώ στην ε, γραμματεία. Η Ελμύρα, Ελμύρες, Λαβύρες, ξέρω εγώ, θα φύγει και θα πάει κάπου αλλού. Θα πάει σε άλλη κοινοβουλευτική ε, επιτροπή. Είχε να χειριστεί σημαντικές εκθέσεις και το πακέτο των σιδηροδρόμων που θα ε, παρουσιάσει βεβαίω και επιτροπολογία, ταχογράφους και άλλα το σχέδιο. Πολύ καλή συνεργάτης υπήρξε, την ευχαριστούμε ιδιαίτερος και για να είμαι και ειλικρινής, πολλοί εκφράζουν τη λύπη τους που ε, φεύγεται. Τότε τι να να συγχαρούμε αυτούς που θα σας πάρουνε, εμείς πάντως στενοχωριόμαστε. Παρ' όλα αυτά σας ευχόμαστε καλή επιτυχία και ε, στην επιτροπή στην οποία θα πάτε. Και νέο πρόσωπο στη γραμματεία

έχουμε στο feedback και τον τριμερή διάλογο. Αυτή η συνάντηση έρχεται και κλεισμένων των ειδών... των